Uh, ladies and gentlemen, I just uh, just a note from the chair to say that the um, there is a gridlock. Κυρίες και κύριοι, ε, υπάρχει πρόβλημα ε, για στο πέρασμα μεταξύ Κομισιόν και εδώ σήμερα το πρωί και η, η Επίτροπος κάπου έχει μπλοκαριστεί εκεί πέρα. Και την περιμένουμε. So, ladies and gentlemen, uh, I think... Um, και κύριοι καλημέρα. Νομίζω τώρα μπορεί να ξεκινήσει και επίσημα η συνεδρίασή μας. Με τα μεγάλης χαράς λοιπόν θέλω να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ και θα ήθελα ιδιαιτέρως να καλωσορίσω την ε, ε, την Επίτροπό μας ε, για τα δικαιώματα των καταναλωτών, η κυρία Κουνέβα, η οποία παρουσιάζεται για τελευταία φορά στην Επιτροπή μας. Έχει εμπλακεί πάρα πολύ στα θέματά μας από όταν ε, καθορίστηκε ως Επίτροπος και παρόλο που ήταν λίγος ο χρόνος μας επηρέασε τόσο πολύ ώστε φαίνεται σαν να είναι εδώ πάρα πολύ καιρό. Ε, το θέμα σας σήμερα είναι η ασφάλεια ε, και φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε να ε, μας, να μας προειδεάσετε και για το τι μέλη γενέστε στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε ευχαρίστω θα σας ακούσουμε. Και σήμερα υπάρχει web streaming, δηλαδή παρουσιάζεται η συνεδρίασή μας εις το διαδίκτυο και η Επίτροπος ήρθε να μας μιλήσει διότι έχει παρακολουθήσει τη δουλειά μας για την εποπτεία της αγοράς και ε, γνωρίζει και ποια είναι τα στρατηγικά μας προγράμματα για την επόμενη πενταετία, για τη δουλειά που σκοπεύουμε να κάνουμε και υπάρχουν και ε, διάφορα άλλα θέματα, ε, η οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων που θα ξανάρθει στα χέρια μας κάποια στιγμή στα επόμενα έτη. Γι' αυτό και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που είστε εδώ η κυρία Επίτροπε και θα μπορέσετε να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. όλους διότι είναι ε, πολύ, ε, πολύ ευχάριστο και, και συγκίνηση για μένα ότι ολοκληρώνουμε την δουλειά της τριετίας και εύχομαι να είστε επιτυχείς και στο μέλλον στη δουλειά μας γιατί ό,τι κάνουμε μετά με, από μια τέτοια εμπειρία με την πολιτική για τους καταναλωτές θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο του σκέπτεστε και στο μέλλον και να ε, παρουσιάζουμε ε, ε, μεγάλες ιδέες όπως είναι η ψηφιακή οικονομία με συγκεκριμένα όμως με συγκεκριμένες προτάσεις που είναι όλες προς όφερος των καταναλωτών διότι πιστεύω ότι οι μεγάλες και μεγαλοσχήμονες ιδέες πρέπει να εξηγούνται στους καταναλωτές με απλά παραδείγματα διότι διαφορετικά είναι υπεροψία να θεωρεί κανείς ότι οι μεγάλες πολιτικές πρέπει μόνο να ενδιαφέρουν την πολιτική ελίτ. Ε, δεν είναι το πνεύμα ούτε της Επιτροπής ούτε του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε ε, να ε, βοηθήσουμε και στην ενεργειακή αγορά και αν οι καταναλωτές δεν αισθάνονται στην τσέπη τους ότι η ολοκλήρωση της ε, είναι καλή ε, για τους ίδιους δεν θα τη στηρίξουν και αν, ε, δεν καταλαβαίνουν κάτι δεν θα το υπερψηφίσουν. Είχα λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Κινέζο Υπουργό όχι για την ε, ασφάλεια του καταναλωτή αλλά για τις εξαγωγές και συζητήσαμε πόσο σημαντικοί είναι οι καταναλωτές και οι οργανώσεις των καταναλωτών. Προσπάθησα δηλαδή να του εξηγήσω πώς δουλεύουμε στην Ευρώπη. Και στο τέλος, αφού είχα ξανλύσει όλα τα επιχειρήματα, του είχα πει «Οι καταναλωτές ψηφίζουν και αυτοί εκλέγουν τους πολιτικούς». Οπότε, ακόμη και από αυτήν την ε, απλοϊκή ε, σκοπιά πρέπει να προσελκύσουμε την κοινή γνώμη, να την ε, έχουμε με το μέρος μας. Ε, αυτό είναι πολύ βασικό για κάθε πολιτικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στις ε, τοπικές κυβερνήσεις. Είναι βασικό να μπορέσει να περάσει μια πολιτική. Γι' αυτό και ξεκίνησα με τις εξηγήσει, γιατί υπάρχουν και άλλες πτυχές. Η οικονομία. Η οικονομία θα ασχοληθεί πολύ περισσότερο με τη λιανική πώληση και το ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά. Το ε, διαδίκτυο έχει ήδη αλλάξει και θα αλλάξει και ακόμη πιο ριζικά τον τρόπο με τον οποίο και παράγουμε και καταναλώνουμε. Οπότε επανέλαβα αυτό το οποίο με είχε εντυπωσιάσει το 2007 όταν προσπαθούσα εναγωνίως να ε, ενημερωθώ και ε, να ε, γνωρίσω τι γίνεται με τις υποθέσεις των καταναλωτών και υπήρχε το άρθρο του Άρθουρ Τόφλερ που έλεγε ότι στον 21ο αιώνα δεν θα υπάρχουν ε, παραγωγής producers και καταναλωτές ε, consumers αλλά prosumers δηλαδή ένα μείγμα των ε, δύο αλλάζουμε απόψε από τη μια μέρα στην άλλη το βλέπετε στο facebook Υπάρχει λοιπόν μια πολύ ε, ενδιαφέρουσα νέα οικονομία, ένας νέος κόσμος, το διαδίκτυο, όλες οι δυνατότητες που διαθέτονται στις υπηρεσίες και στα προϊόντα. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Δεν πρέπει δηλαδή να πετάξουμε τις παλιές ε, πολιτικές, την ασφάλεια και τα ασφαλή προϊόντα, αλλά να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις για την ε, συνολική ασφάλεια γιατί η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στις επάλξεις και να ηγείται και είναι ο καλύτερος τρόπος μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις κυβερνήσεις μας. Μπορούμε να εξάγουμε καλύτερα τα προϊόντα μας, μπορούμε να τους εξηγήσουμε πώς φτάσαμε σε αυτά τα συμπεράσματα μετά από επίπονη εργασία, δεκαετίες ε, στη σειρά και πώς ε, εφαρμόζουμε την καλή διακυβέρνηση. Αυτή είναι η δύναμή μας και για την αγορά. Η φωνή μας ε, ε, πολλαπλασιάζεται από εκατομμύρια καταναλωτών. Πάντοτε λέγω και όταν ήρθα και σας είδα και γύρισα στον Μάλκολμ και του είπα ότι αυτή είναι η επιτροπή μου, είμαι η επιτροπό σας. Πάντοτε θα με ακολουθεί η σκέψη από τη σκοπιά του καταναλωτή, διότι πιστεύω σε αυτή την πολιτική, πιστεύω στην επιτροπή σας, είμαι ε, πολύ ευτυχής ε, αν έχετε έξυπνες ιδέες ή ε, διάφορες εκδηλώσεις να σας ακούσω και να εμπνέομαι από τη σοφία σας. Και μία τελευταία φράση. Θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων και των επιτροπών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρώπη. Εάν μιλάμε για τον 21ο ε, αιώνα που συνδυάζει την παραγωγή με την κατανάλωση από την πλευρά της διακυβέρνησης, από τη διατύπωση των πολιτικών θα πρέπει να προέχει η συμφωνία. Όσο πιο ενωμένοι είμαστε τόσο καλύτερα θα αποδίδουμε. Πρέπει να συμφωνήσουμε για, περί του πρακτέου και ε, περί των τρόπων με τον οποίο θα επιτύχουμε τις επόμενες φάσεις. Αυτή η Επιτροπή λοιπόν θα έχει έναν εξαιρετικό ρόλο για να ε, εργαστεί ε, σε συνεργασία με τις επιτροπές και τις πολιτικές ομάδες στο μέλλον. Ε, συνάντησα εχθές τον κύριο Ντάλι, τον νέο επίτροπο, ο οποίος είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα και αυτό είναι πολύ βασικό, διότι η εφαρμογή και η διεκπαιρέωση των παραπώνων είναι έχουν μπει ήδη σε μια σειρά. Άρα ελπίζω ότι και στο μέλλον θα μπορείτε να υποφεληθείτε από αυτόν τον τομέα τον οποίο εξετάζουμε και το καλύτερο για μένα που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας είναι ότι είμαι στην Επιτροπή μου με ε, τους ομολόγους μου. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε τώρα με την εργασία μας. Τα όσα σας είπα για την ε, εργασία μου κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να σας ευχαριστήσω για τα συγκεκριμένα θέματα, για την εποπτεία της αγοράς στο πλαίσιο της ε, γενικής ασφάλειας των προϊόντων. Αυτό είναι το επόμενο βήμα Ήσασταν μεγάλοι υποστηριχτέ για την πολιτική κατανάλωτη και για τις προσπάθειες της τοποθέτησης πολιτικής αυτής στην καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτικών γενικότερα. Και πάλι στον τομέα της εποπτείας της αγοράς και την ασφάλεια των προϊόντων, πραγματικά με τη διαφορά. Ε, θα ξεκινήσω λέγοντας, ε, μιλώντας για κάτι που θεωρώ ήταν ένα από τα καθοριστικά σημεία κατά την ε, θητεία μου ως Επιτρόπο. Το 2007 είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν από τους μεγαλύτερους γρίφους, όπου 20 εκατομμύρια παιδιά, παιχνίδια αφαιρέθηκαν από τα ράφια. Αυτό κατέληξε στην απώλεια της εμπιστοσύνης ε, των καταναλωτών η οποία θα πρέπει να αποτελεί μια σταθερά της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς αλλά και της παγκόσμιας αγοράς. Φαντάζομαι πως όλοι μας εδώ θέλουμε περαιτέρω να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά, θέλουμε οι επιχειρήσεις μας να εξακολουθήσουν να υποφελούνται από τις παγκόσμιες ε, αλυσίδες παροχής, και να κινητοποιούμε την παγκόσμια ανάπτυξη. Αφού θέλουμε αυτό το πράγμα, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι πω οι καταναλωτές θα εμπιστεύονται τα προϊόντα που αγοράζουν και τι υπηρεσίε που χρησιμοποιούν ακόμα περισσότερο όταν προέρχονται από μια ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό θεώρησα ότι έπρεπε να αντιδράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά να διασφαλίσουμε όχι μόνο ότι τα ανασφαλή προϊόντα θα έβγαιναν από την κυκλοφορία όσο γινόταν πιο γρήγορα, αλλά και να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να συμβούν παρόμοια πράγματα και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Κάτι τέτοιο χρειάζεται πολλά και διάφορα μέτρα, καθώς και συνεχή προσοχή. Δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την νομοθεσία. Άρα λοιπόν τι κάναμε, επιμείναμε τα κράτη-μέλη να αυξήσουν την υποπτία τους. Ξεκινήσαμε με προγράμματα για να δούμε για την ασφάλεια του, των παιχνιδιών και πείσαμε τον τομέα τον κλάδο της κατασκευής παιχνιδιών να επιμείνουν για την ασφάλεια. Πίεσαμε επίσης τις κινέζικες αρχές να επιμείνουν για τους ελέγχους εξα... στους εξαγωγείς τους και ε, ξεκινήσαμε μαζί με τους Αμερικανούς ομολόγους μας ε, να ανταλλάσσουμε εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη. Ωστόσο, το να υπάρχει για το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό και προϋπόθεση όπως δείχνει και η αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας. Μετά από το καλοκαίρι εξετάσαμε το ευρύτερο πλαίσιο για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με το πακέτο που θα ξεκινήσει να ισχύει τον Ιανουάριο, να αρμονίσαμε και ενισχύσαμε τις ε, προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις αλλά και για τις αρμόδιες αρχές. Και, και τώρα για τις γενικές αρχές. Ε, το σύστημα αυτό εκτιμήθηκε γρήγορα και έδειξε πως ήταν ένα ισχυρό μέσο για τη διασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου ασφάλειας του καταναλωτή. Ένα πρότυπο το οποίο επεκτείνεται και στα μη καταναλωτικά προϊόντα και σε άλλα είδη κινδύνων και που θεωρείται ως υπόδειγμα από πολλές χώρες ε, εκτός Ένωσης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να επαναπαυτούμε στις δάφνες μας. Πάντοτε έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέες εξελίξεις, όπως η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η τεχνολογία, οι μεγάλες μετακινήσεις στις μεγάλες και αλλαγές στις μεγάλες αλυσίδες ε, παροχής. Αυτό θα πρέπει να μας αναγκάζει να αντιδρούμε γρήγορα στις, στις συνεχείς αλλαγές στον χώρο της αγοράς. Και γι' αυτό και αρχίσαμε ήδη να, αντιδρα... να αναθεωρούμε την οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων που ισχύει εδώ και έξι χρόνια τώρα στη μορφή αυτή που έχει. Πρέπει λοιπόν τι μελλοντικέ προκλήσει να τι ε, αντιμετωπίσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, θα θέλαμε να εστιάσουμε σε σαφέστερου ε, κανόνε για την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων και πολλέ φορέ μου ζητήσατε να το κάνω αυτό λιγότερο η ε, γραφειοκρατική διαδικασία της τυποποίησης και περισσότερη ευελιξία στην εφαρμογή των ε, μέτρων έκτακτη ανάγκης. Η δική σας υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επόμενης νομοθετικής διαδικασία, της επερχόμενης μάλλον νομοθετική διαδικασία, θα είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, ε, όλα αυτά τα μέτρα, ακόμα και αν είναι τέλεια, δεν θα χρησιμεύσουν αν δεν είναι εφαρμοστούν σωστά. Πράγμα το οποίο με οδηγεί στην εποπτεία της αγοράς. Τα, πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια από 140 μόνο το 2003 ήρθαμε, ανεβήκαμε στη 100, στις, ε, στα 1850 μέτρα. Αυτή η ανάπτυξη δεν ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται μόνο στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, είναι περισσότερο δέσμευση από αυτούς που ασχολούνται με την ασφάλεια των προϊόντων, την εταιρεία και τις ε, αρμόδιες αρχές. Η ευθύνη για την εμπορία ασφαλών προϊόντων σαφώ βαραίνει μόνο τι επιχειρήσει. Κανένα δεν πρόκειται να, την, να, να, να αφαιρέσει μάλλον την ευθύνη από εκείνου. Ωστόσο, ταυτόχρονα χρειάζεται να υπάρχει αξιόπιστη προσπάθεια επιβολή. Δυστυχώς ορισμένοι φορεί δεν είναι πάντοτε σε θέση να ελέγξουν τους κινδύνους για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. Και ακόμα χειρότερο, ορισμένοι άνθρωποι ακολουθούν μόνο τους κανόνες μόνο όταν υπάρχει περίπτωση να τους πιάσουν. Και γι' αυτό και η εποπτεία της αγοράς είναι τόσο σημαντικό ζήτημα, όχι μόνο για να προστατευτούν οι άνθρωποι, οι καταναλωτές από τα μη ασφαλή προϊόντα, αλλά και για να υπάρχει ισότιμο πεδίο για τις ε, επιχειρήσεις. Θα ήθελα να τονίσω ότι η εποπτεία της αγοράς αντιμετωπίζει όχι μόνο χρηματοπιστωτικές προκλήσεις μετά από την κρίση, αλλά και το θέμα της ε, συνεχιζόμενης παγκοσμιοποίησης με όλο και περισσότερα προϊόντα που μπαίνουν στην εσωτερική αγορά της Ένωσης από τρίτες χώρες, καθίσταται όλο και πιο δύσκολο το να εφαρμοστεί μια απλά εθνική προσέγγιση στην επιβολή. Εγώ βλέπω πως ε, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αρχών και μεταξύ, με τους διεθνείς μας ομολόγους. Καταρχήν, ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Αρχές Εποπτείας. Η φύση της αγοράς μας, ε, συνδυασμένη με τις παγκόσμιες αλλαγές, ε, καθιστά απαραίτητη την δημιουργία μιας, ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών. Και γι' αυτό και η Κομισιόν έχει κάνει πρόταση για συντονισμό ε, των δραστηριοτήτων των κρατών μελών, κυρίως μέσω της οικονομικής αρρωγής για κοινέ δράσεις. Για παράδειγμα, τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουμε υποστηρίξει το ΠΡΟΣΕ, ένα δίκτυο που συγκεντρώνει τις αρχές εποπτείας της αγοράς στα κράτη-μέλη. Ε, για την ανάπτυξη των καλύτερων πρακτικών και για την ενίσχυση του συντονισμού. Οι δραστηριότητε του ήδη έχουν καταλήξει σε σημαντικές ε, βελτιώσεις ε, στη λειτουργία στα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των τελωνιακών αρχών. Και αυτό βασικά χάρη στην υποστήριξή μας που το ΠΡΟΣΕ θεωρείται ως το de facto όργανο συντονισμό για την ευρωπαϊκή εποπτεία της αγοράς. Ε, με χαρά θα σας εξηγήσουν τις δραστηριότητες τους, αν το επιθυμείτε. Επίσης, έχουμε δώσει επιχορηγήσεις για συγκεκριμένες δράσεις, για τα παιχνίδια, για τους εξοπλισμούς στις παιδικές χαρές, τα χριστουγεννιάτικα φώτα και τους αναπτήρες. Αυτέ οι δράσει δίνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Χθε, για παράδειγμα, συναντήσαμε εκπροσώπου των κρατών μελών και ε, είδαμε τα αποτελέσματα κοινών δράσεων. Ε, για τα ε, για τα συγκεκριμένα τους εξοπλισμούς των για τα σολάριουμ. Ε, είδαμε πως υπάρχουν ε, ακόμα, ξεπερνώνται τα επίπεδα ε, ραδιενέργειας σε πολλές περιπτώσεις και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν προσαρμογές. Οι προσπάθειες της εποπτείας σε πολύ μεγάλο βαθμό κατευθύνονται από τις εθνικές προτεραιότητες και πρακτικές και παραμένουμε διχασμένοι στην ε, ενιαία μας αγορά. Η αξιολόγηση κινδύνων για τα ίδια προϊόντα αποκλίνουν παρά τις κοινέ κατευθυντήριες γραμμές. Επίσης, όλα αυτά είναι διαπραγματικότητα όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα και τις ποινές. Η ανάμειξη των τελωνιακών αρχών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προθυμία τους σε εθνικό επίπεδο να ασχοληθούν με τα θέματα της ασφάλειας των προϊόντων. Η επιτυχής αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων θα απατήσει μια αλλαγή σημαντική και ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στα κρατη Χρειάζεται μια, ένα πραγματικό δίκτυο ευρωπαϊκό για την εποπτεία που να μπορεί να προσαρμοστεί και να μπορεί να θεσπίσει τις ε, ευρωπαϊκές προτεραιότητες επιβολής. Ένα τέτοιο δίκτυο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις τελωνιακές αρχές ώστε να υπάρχουν περισσότερα και πιο αποτελεσματικά σημεία ελέγχων. Η εμπειρογνωμοσύνη θα πρέπει να γίνεται ε, κοινό κτήμα με περισσότερη γενεδορία και με περισσότερη αποτελεσματικότητα. Χωρίς κάτι τέτοιο... Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι σαν να ψάχνουμε βελόνες τάχυρα. Χρειάζεται δε η επιβολή να γίνεται πιο, πιο κοντά στην πηγή, ώστε να μην πνιγούμε στον όγκο των προϊόντων που προέρχονται από τη διεθνή αγορά. Και έτσι έρχομαι και στους διεθνούς μας, ε, διεθνείς μας εταίρους, που, χρειάζεται και μια διεθνής αρχή για την επιβολή κοινών κανόνων. Και γι' αυτό εξ αρχής της εντολής μου, εγώ ανέπτυξα στενότερους δεσμούς με τους διεθνούς μας εταίρους, είπα Κίνα μεταξύ αυτών. Έχουμε εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διαπραγματευτούμε συμφωνία με τους Αμερικανούς ομολόγους μας, ε, να ανταλλάζουμε πληροφορίες για τα επικίνδυνα προϊόντα, τα ατυχήματα λόγω μη ασφαλών προϊόντων, ε, αξιολογήσεις κινδύνου. Οι κοινέ πληροφορίες θα πρέπει να βελτιώσουν την δυνατότητά μας να προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους καταναλωτές και με την Κίνα τώρα. Επίσης εξετάζουμε περαιτέρω τρόπους για την ενίσχυση της συνεργασίας μας. μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προτινόμενες προσεγγίσεις είναι αυτό που εγώ αποκαλώ η εποπτεία άνευ συνόρων, όπως με το, το, τα σύνορα. Δηλαδή, η έλεγχη των εξαγωγών από, την Κινέζικη αρχή, από τις Κινέζικες αρχές θα πρέπει να συνοδεύονται από ελέγχους και από τις Ευρωπαϊκές αρχές, έτσι ώστε να έχουμε μια προσέγγιση εποπτείας από το εργοστάσιο μέχρι την πόρτα του καταναλωτή. Ε, θα μπορούμε έτσι να, να χειριστούμε τα προβλήματα στην πηγή τους. Και γι' αυτό όχι μόνο θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει επαφέ με τους εταίρου μας, μάλιστα τον Νοέμβριο του 2008 συγκεντρώσαμε, μάλλον συγκαλέσαμε μια συνάντηση Αμερικανών και Κινέζων ε, εκπροσώπων για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ελπίζω πως αυτή η τριμερή συνεργασία θα συνεχιστεί, γιατί φάνηκε πως ήταν μια πολύ χρήσιμη, ένα πολύ χρήσιμο βήμα για τη διάδοση των ιδεών και για την ανάληψη πολιτικών δεσμεύσεων για τις περαιτέρω δράσεις. Επίσης, συμμετέχουμε στον ΟΣΑ και στο Διεθνές ε, Συμβούλιο για την Προστασία του Καναλωτή, ώστε να προσχωρήσουμε και σε πολυμερές πλαίσιο. Και πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να τονίσω ότι όπως και η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα και η συντονισμένη προσέγγιση στην εποπτεία των αγορών δεν θα συμβεί εν μία νυχτή. Θα χρειαστεί σημαντική προσπάθεια και επιμονή από όλους τους εμπλεκόμενους μεταξύ των οποίων είναι και δική σας η Επιτροπή και από καθέναν από εσάς μεμονωμένα. Θα μπορέσουμε να έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ενιαίο νομοθετικό αποτελεσματικό πλαίσιο για την παγκόσμια προστασία που θα προστατεύσει τους Ευρωπαίους ε, καταναλωτές τα επόμενα χρόνια και μόνο όταν ο καταναλωτής αποκαταστεί στην εμπιστοσύνη του στα προϊόντα και στην ασφάλειά τους ε, θα είναι ε, και είναι πολύ μεγάλο το καθήκον αυτό. Είναι 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες σε πολύ, πολύ σπουδαίο και ευγενέ καθήκον. Μύρισα πάρα πολύ γρήγορα, όσο μπορούσα πιο γρήγορα για να τελειώσω στην ώρα μου. Και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Επίτροπε, για την ιδιαίτερα ε, περιεκτική και ε, στρατηγικού τύπου παρουσίαση ε, που μας κάνατε. Νομίζω ότι η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει την εργασία της σε αυτό τον τομέα και νομίζω ότι ε, όσον αφορά την ταχύτατη αντίδραση έναντι των κινέζικων αρχών, ε, νομίζω ότι μπορέσατε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες ε, διεθνούς συνεργασίας. Και από αυτό θα αποφοληθούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, αλλά και καταναλωτές ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω ότι η διεθνή συνεργασία μπορεί να συνεχίσει και ήδη υπάρχει κάποια προσέγγιση εκ μέρους των ΗΠΑ και στην Κίνα είχαμε μια ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα επίσκεψη στη Σανγκάη ως συνέχεια των εργασιών σας. Η κυρία Γκέπαρτ είναι ιδιαίτερως ε, δραστήρια εντό της κινέζικης ε, αντιπροσωπείας και νομίζω ότι μπορούμε να ε, ασχοληθούμε περισσότερο με τη δουλειά μας εδώ, γιατί τα μέλη των αντιπροσωπιών πραγματικά κάνουν σημαντική δουλειά. νομίζω μας αφήσετε μια πολύ σημαντική κληρονομιά. Και ε, πραγματικά ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να ακούσουμε τα όσα έχετε να πείτε σχετικά με τα φώτα των ε, Χριστουγέννων. Οι συνάδελφοι προετοιμάζουν ήδη τις ανακοινώσεις ε, τύπου προκειμένου να προλάβουν κάποια σοκ εκ μέρους των Ευρωπαίων καταναλωτών σε σχέση με τα Χριστούγεννα, γιατί είναι πραγματικά διάσημες οι ρίσεις σας. Τώρα, θα δώσω το λόγο στους συντονιστές, τον κύριο Σβάπ, την κυρία Κέπαρτ, τον κύριο Κρότσμαν, δεν ξέρω, την κυρία Φιλίππη. την κυρία Σαλτεμόζε, την κυρία Στάιλερ κλπ. Right. Right. Let's start then with Mr. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Σουάπο. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Ε, δεν πειράζει αν αρχίσει αργότερα η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητή Επίτροπε, αγαπητή κυρία Κούνεβα. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ που ακόμα και σε αυτή τη μεταβατική περίοδο μεταξύ της παλαιάς εντό και νέας ε, επιτροπής ε, εξακολουθεί να παίρνει σοβαρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι για την εκ μέρους του ΕΛΚ μπορούμε να πούμε ότι κατά τη διάρκεια ολόκληρης της θητείας σας ε, πραγματικά είστε ιδιαίτερα δραστήρια και πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη χαρά για μας να συζητούμε μαζί σας. Έστω και αν είχαμε διαφορετικές θέσεις, πάντοτε ήταν ξεκάθαρο ότι εσείς θέλετε να πάτε προς τα μπρος. Θέλετε να ανοίξετε το δρόμο προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση από από 27 ισότιμες χώρες. Αυτό ωφέλει ιδιαίτερα ιδιαίτερες εργασίες μας και νομίζω ότι αυτό σας ε, διαφοροποίησε από τους συναδέλφους σας. Στα εισαγωγικά σας σχόλια μιλήσετε για την, το συνδυασμό μεταξύ ε, καταναλωτών και επιχειρήσεων και επιχειρηματιών και αυτό αφορά εμάς, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ε, ελεύθερης αγοράς, γιατί οι καταναλωτές συμμετέχουν σε μια αγορά, εντός της οποίας οι επιχειρηματίες δεν έχουν τον ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν. Και νομίζω ότι εδώ πραγματικά δώσετε το σωστό τόνο. Αυτό δεν το κάνετε μόνο στο παρελθόν όσον αφορά τα παιχνίδια από την Κίνα, όπου πραγματικά ε, μπορέσετε να παρέμβετε ιδιαίτερως αποφασιστικά και με την ε, επιτυχία. Ε, αλλά είδαμε και ότι στην οδηγία για τα παιχνίδια, η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων όσον αφορά την ε, καταναλωτική πολιτική, ε, πάντοτε ε, συνοδευόταν από κάποιες τριβές και προβλήματα. Και νομίζω ότι η χθεσινή απόφαση ότι θα γραφεί στον πρόεδρο τη Επιτροπή μια επιστολή ούτω ώστε και μελλοντικά η καταναλωτική πολιτική να μπορέσει να συντονίζεται αποτελεσματικά ούτω ώστε να έχει έναν ενιαίο χαρακτήρα και να μην είναι κατακαιρματισμένη σε πολλέ γενικέ διευθύνσει. Αυτό το οφείλουμε σε εσά κυρία Κούνεβα. Τέλο, όσον αφορά τη σημαντική σα πρόταση για την ανάπτυξη των δικαιωμάτων καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, θα ήθελα να πω ότι δεν ήταν μια απλή απόφαση για εσά να υποβάλλετε την πρόταση αυτή στη βάση τη αρχή τη πλήρου εναρμόνιση. Με τους σκιώδεις συγητές, ως συγητής, εγώ προσπαθώ να επιλύσω τα προ... δυσεπίλητα προβλήματα στον τομέα αυτό και να εξαύρω κάποιες λύσεις. Αλλά βασικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που κάνετε αυτό το βήμα προς τα μπρος, γιατί όσον αφορά την εσωτερική αγορά νομίζω ότι με τέτοιου είδου προτάσεις προωθείται αυτή η υπόθεση. Και χρειαζόμαστε περισσότερους υπέρμαχους της εσωτερικής αγοράς. Εσείς είσαστε μια βασική υπέρμαχος της εσωτερική αγοράς και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σα ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κούνε. Äh, Και νομίζω ότι μας δείξατε πόσο ε, σοβαρά παίρνετε το ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών. Ε, και γι' αυτό ως ε, σοσιαλδημοκράτες και δημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά θα θέλαμε να σας αποτίσουμε φόρο τιμής, διότι δεν είναι αυτονόητο όπως ε, μας έχει δείξει πείρα μας από την συνεργασία με άλλους επιτρόπους που στο τέλος της θεία τους εξαφανίστηκαν. Θα θέλαμε λοιπόν να σας πενέσουμε και να σας πούμε ότι ακόμα και εντός της δικής μας πολιτικής ομάδας δεν, υπήρχαν, ε, δεν υπήρχε πάντοτε ομοφωνία. Παρ' όλα αυτά η καλή συνεργασία ήταν σημαντική, υπήρχε διαφάνεια, ε, υψηλός βαθμός διαφάνειας και ειλικρίνεια. Αλλά υπάρχει ένα σημείο όπου εδώ δεν είμαστε απολύτως σύμφωνοι. Αφορά στην ε, προσέγγιση από πολιτική άποψη όσον αφορά την σημασία της προστασίας των καταναλωτών. Γιατί είπατε μόλις προηγουμένως στα εισαγωγικά σας σχόλια όσον αφορά την παρακολούθηση της αγοράς ότι η προστασία των καταναλωτών είναι ακρογωνίως λήθος για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Και εμείς οι Δημοκράτες λέμε όχι, ε, ισχύει ακριβώ το αντίθετο. Η εσωτερική αγορά είναι για τους καταναλωτές. Κάνουμε μια πολιτική υπέρ των πολιτών και όχι για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι μια φιλοσοφία ε, που εμείς και η Κομισιόν ε, δεν είμαστε πάντοτε σύμφωνοι. Ωστόσο, θα πρέπει να σε επανέσουμε το γεγονό ότι έχει υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τον γεγονό ότι ο καταναλωτή χρήζει προστασία και δεν ε, εξισώνεται με φτηνή ε, προσφορά ή δεν τον προσελκύουμε με τη φτηνή προσφορά, αλλά χρειαζόμαστε μια προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας. Κάτι το οποίο σηματοδοτεί πραγματικά μια καμπή στην πολιτική αυτή. Τώρα, όσον αφορά την παρακολούθηση τη αγορά, αναφέρεται κάποια σημεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά αναφερθήκατε στην ανιχνευσιμότητα των προϊόντων, ούτω ώστε να μπορεί κανείς να προσεγγίσει τα προβλήματα στη ρίζα τους και όχι να προσπαθεί να τα επιδιορθώσει εκ των υστέρων. Και ένα άλλο θέμα που εντάσσεται εδώ, ε, κάτι παραλείψετε κατά την άποψή μου, ε, το πρόβλημα της ε, σήμανσης ασφαλείας ως προέλευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θα πρέπει να συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα ασφαλείας. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε με τον νέο Επίτροπο. Αναφερθήκατε στο θέμα της ασφάλειας της υπηρεσίας. Νομίζω ότι εδώ ε, χρειάζεται να γίνουν κάποια πράγματα. Όσον αφορά τα προϊόντα έχουμε ε, προχωρήσει αρκετά, έστω και αν η παρακολούθηση της αγοράς παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Αλλά όσον αφορά τις υπηρεσίες και εδώ με αυτό εννοώ τις οικονομικές υπηρεσίες, για παράδειγμα τις μικρο... Ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή για τα ε, αγοραστικά κέντρα ε, αυτή είναι το τομεί όπου χρειάζεται να γίνουν κάποια πράγματα, όπου υπάρχει πραγματικά ένα ευρύ πεδίο, ευρύ φάσμα προβλημάτων, τα οποία καλούμεθα να προσεγγίσουμε. Τελευταίο σημείο. Ε, θα είχα να πω και άλλα πράγματα, αλλά θέλω να θέσω το χρόνο στου συναδέλφου. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν διαφορέ όσον αφορά την ε, προσέγγιση τη οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Εμεί, οι σοσιαλδημοκράτε, λέμε ξεκάθαρα ότι αυτή η προσέγγιση της πλήρους εναρμόνισης δεν μας βρίσκει σύμφωνος, δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε. Για μας είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε και ότι θα πρέπει ε, να έχουμε ένα σύστημα ελάχιστης εναρμόνισης ε, ή δυνατόν υψηλό επίπεδο. Αλλά παρόλα αυτά να υπάρχει δυνατότητα για τις χώρες μέλη ενδεχομένως να εφαρμόζουν ε, εν μέρη καλύτερες επιμέρους ρυθμίσεις. Αναφέρεται η ίδια στην αρχή της παρουσίασής σας τα πολλά προϊόντα και τις πολλές υπηρεσίες που φτάνουν στην αγορά που δεν είναι δυνατόν να ε, κοπούν στα μέτρα μιας ε, οδηγίας. Ε, και στο πλαίσιο της, οδηγίας, της εργασίας αυτής δεν μπορούμε να παρακολύσουμε το έργο των διαφόρων οργανώσεων για την προστασία των καταναλωτών. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το στηρίξουμε όπως σας είπα. Έχω τον κύριο ε, Κρόετσμαν, στη συνέχεια τον κύριο Τρενταφυλλίδη και μετά θα περάσουμε στους άλλους ομιλητές. Ο κύριος Κρόετσμαν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κυρία Κούνεβα. Στην ομιλία σας δείξατε ότι η παρακολούθηση της αγοράς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Μία προστασία των καταναλωτών χωρίς την παρακολούθηση της αγοράς μπορείτε να την ξεχάσετε απλούστατα. Αυτό είναι το α και το μεγα. Είπατε, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της βιομηχανίας των παιχνιδιών, ότι εκεί υπάρχουν εκατομμύρια εισαγωγών ε, προς την Ευρώπη. Και βεβαίως ανακύπτει το ερώτημα πώς μπορεί να λειτουργεί αυτή η παρακολούθηση της αγοράς. Είπατε ότι υπάρχει μια παγκόσμια εργασία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια παγκόσμια προστασία. Ε, και συνεπώς θα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια να συνεργαστούμε με τις εξαγωγικές χώρες, αλλά ταυτόχρονα και να προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τις σύγχρονες δυνατότητες είτε μέσω του σκάνινγκ είτε μέσω των microchips ούτως ε, ώστε εκεί όπου παράγονται τα προϊόντα αυτά και με τη βοήθεια κάποιων δειγμάτων να έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια επαρκή σήμανση ούτως ώστε όταν τα προϊόντα αυτά εισάγονται στην Ευρώπη να μπορούν να παρακολουθούνται. Και το ίδιο βεβαίως ισχύει και για την παρακολούθηση της αγοράς παγκοσμίω Έχουμε διάφορους ε, λιμένες στην Ευρώπη όπου φτάνουν ε, πάρα πολλές αγωγές, το Αμβούργο, το Ρότερνταμ, η Γένοβα κλπ. Για παράδειγμα, εκεί είναι δύσκολη βεβαίως η παρακολούθηση αλλά είπατε ότι πρέπει να υπάρχει μια δικτύωση. Πρέπει να υπάρχει ένα παγκόσμιο δίκτυο εκεί όπου παράγεται, όπου, ε, στον πρώτο παραγωγής, αλλά και στην Ευρώπη. Ε, αυτό είναι σημαντικό και δεν ισχύει μόνο για την βιομηχανία των παιχνιδιών, αλλά και για τα ζυζανιοκτώνα ή για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ε, ζυζανιοκτώνα ε, και εντομοκτώνα ε, και όπου υπάρχουν μαζικές ε, παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Ε, έξω και η παράκλησή μας, το θέμα της παρακολούθησης της αγοράς να συμπεριληφθεί και στη μέση διάταξη των επόμενων πέντε ετών. Το εξαγγείλετε άλλωστε στην ομιλία σας. Είπατε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα σύγχρονα μέσα, ούτως ώστε, ε, τα ψηφικά μέσα, ούτως ώστε να μπορούν να παρακολουθούνται αυτά τα ε, εισαγόμενα προϊόντα. Και βεβαίως στο πλαίσιο της επίδειξης μιας ελληνικής προς τις χώρες που έχουν εξαγωγικούς, εισαγωγικούς λιμένες. Και ε, βεβαίως είναι, ξέρετε για παράδειγμα ότι στη Γερμανία ε, η παρακολούθηση γίνεται από τα ομόσπαντα κρατήδια και ο έλεγχος αυτός ε, στα λιμάνια είναι δυσχερής. Θα πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε αλληλεγγύη και να προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη δικτύωση, ούτω ώστε να προχωρήσει η υπόθεση αυτή εις όφελος της εσωτερικής αγοράς, αλλά και της προστασίας των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τρενταφυλλίδης. Ήθελα να συμφωνήσω με τα σχόλια της κυρίας ε, Κέπαρτ ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να εργάζεται πάντοτε υπέρ του καταναλωτή στη δική μας ε, συνεισφορά, τη συνεισφορά της δικής μου πολιτικής ομάδας, της εργασίας της Επιτροπής μας, πάντοτε έχουμε σαν αφετηρία της, ε, των προτάσεων που κάνουμε το ερώτημα πώς μπορούν τα συμφέροντα του καταναλωτή να προστατευτούν και να ενδυναμωθούν περισσότερο. Από αυτό το φαγό καλωσορίζουμε τα όσα μας έχει πει η Επίτροπος για την εποπτεία της αγοράς και με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση της πολιτικής μου ομάδας προς το πρόσωπο της Επιτρόπου και να της ευχηθώ τα καλύτερα στο νέο της πόστο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους συναδέλφους οι οποίοι ήρθαν ε, για τις 10 <clears throat> και ε, να σας πω ότι αργήσαμε να ξεκινήσουμε γιατί η κυρία Επίτροπος είχε μπλέξει στην κίνηση αλλά θα σας παρακαλούσα αν έχετε συζητήσεις να τις κάνετε εκτός εθούσης. Θα αρχίσουν οι ψηφοφορίες γύρω στις 10 και 4. Δηλαδή αν υπεύθυνοι πολιτικών ομάδων ψάχνουν ακόμη τα μέλη τους έχουν ένα τέταρτο να τους βρουν και να τους προσκομίσουν. Έχουμε διάφορες παρεμβάσεις ακόμη και παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί ναι μεν είμαι χαλαρός αλλά δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Η κυρία Σόλτερ Μόζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα προσπαθήσω να πω στην κυρία Κούνεβα ότι βεβαίως και εγώ θα ήθελα να του ευχηθώ κάθε επιτυχία για το μέλλον και να την ευχαριστήσω που ήταν διαθέσιμη στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής και ανοιχτή στο διάλογο. Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με αυτά που είπατε σχετικά με την εποπτεία της αγοράς, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα και είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουμε αυτό το οποίο και εσείς ε, ε, επιζητάτε διότι ε, πριν από ένα χρόνο υιοθετήσαμε το Good Package, το πακέτο για τα εμπορεύματα και αναθεωρήσαμε και την ε, νομοθεσία για την εποπτεία της αγοράς και τα κράτη-μέλη πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστούν στα θέματα εποπτείας της αγοράς. Και πριν από ένα-ενάμιση μήνα στην Επιτροπή μας προσπαθήσαμε να δούμε πόσο έχουν προχωρήσει τα κράτη-μέλη. Είδαμε λοιπόν ότι μόνο δύο κράτη, η Κύπρος και η Δανία, είχαν διαθέσει περισσότερους πόρους για την εποπτεία της αγοράς. Όταν λοιπόν κοιτάμε την νομοθεσία, όταν την αναθεωρούμε και θέλουμε να την καταστήσουμε πιο αυστηρή, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε ανταπόκριση από τα κράτη-μέλη και απέχουμε ακόμη πάρα πολύ από μια κατάσταση όπου θα είχαμε στην εσωτερική αγορά ασφαλή προϊόντα. Μας είπατε ότι θα θέλατε να υπάρχει μια πιο στενή συνεργασία. Βλέπετε ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας και θα πρέπει να πιέσουμε τα κράτη-μέλη και ελπίζω ότι αυτό θα κάνει και η Επιτροπή στο μέλλον. Ευχαριστώ. Θέλω επίσης κυρία Σάλτε Μόζαρ να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά σας ε, στο θέμα της ε, εποπτείας αγοράς. Με συγχωρείτε. Έχουμε την κυρία Στάιλερ και την κυρία Βάιλερ, ε, με συγχωρείτε αλλά εννοούσα την κυρία Βάιλερ πρώτα. Δεν πειράζει, αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Αλλά είναι καλό κύριε Πρόεδρε που μιλώ μετά τη συνάδελφο Σάντε Μόζερ διότι και εγώ θέλω να προσθέσω στην εποπτεία της αγοράς. Αλλά καταρχήν κυρία Επίτροπε και από μένα ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ε, όντως η Επιτροπή σας, είμαστε η Επιτροπή σας, είστε η Επίτροπό μας, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Τώρα έχουμε πέντε και δεν ξέρουμε ε, ποιος θα είναι υπεύθυνο γιατί. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να σας πω ότι ήθελα να αναπτύξω το θέμα του scoreboard για τους καταναλωτές, του πίνακα βαθμολογίας και το, συζητάμε, ε, το συζητήσαμε χθε εκτενώς. Εσείς ήσασταν η πρώτη η οποία το είχε παρουσιάσει κατόπιν προτάσεώς μου και ε, αντιδράστε πολύ γρήγορα. Δεν είναι συνηθισμένο ε, επίτροποι να αντιδρούν τόσο γρήγορα στις επιθυμίες των ε, ευρωβουλευτών. Αλλά ε, διαπιστώνω από την άλλη πλευρά ότι οι εθνικές ε, εποπτικές αρχές έχουν βελτιωθεί και με τα τελωνία, αλλά παραδείγματος χάρη διαπιστώνω ότι έχουμε τόσα προβλήματα με τα φωτάκια για τα δέντρα τώρα. Ε, για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ε, βλέπω ότι αναφέρετε στην ιστοσελίδα σας τι κατακρίνεται στο δίκτυο διανομής και στα διάφορα κράτη, αλλά γιατί υπάρχουν ε, τόσες ελλείψεις, γιατί η παραγωγή των φώτων αυτών έχει ξεκινήσει από το Φεβρουάριο-Μάρτιο, δηλαδή έχει προετοιμαστεί πολύ καιρό. Μπορείτε να μας πείτε κάτι, γιατί τώρα πια είναι αργά. Δηλαδή πάρα πολλοί ε, πολίτες ε, και ε, δημοτικές αρχές έχουν ήδη κρεμάσει τις γερλάντες οι οποίες φωτίζουν και μας λέτε ότι μπορεί να υπάρξουν υπερθερμάνσεις και κρίξεις και νομίζω ότι είναι αργά πια τώρα για να το επισημάνει κανείς. Η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε ε, καταρχήν θα ήθελα προσωπικά να σας ευχαριστήσω για την ειλικρίνειά σας. Πάντοτε απαντούσατε στα ερωτήματά μας και θα είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσει κανείς το άτομό σας αυτή τη θέση ε, διότι έχετε ασχοληθεί με όλα τα θέματα. Σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας ε, για τα αρκουδάκια στην κάθη στο Αμπερντίν και ίσως ε, θα ήθελα να μας διευκρινίσετε και να μας ε, ε, καθησυχάσετε ότι αυτά τα αρκουδάκια έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Επίσης πριν από μερικές μέρες ε, μας στείλατε ένα έγγραφο το οποίο είναι τρομακτικό. Προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους να μην χρησιμοποιούν αυτά τα sunbeds, τα στρώματα για ηλιοθεραπεία, αλλά ε, ελπίζω ότι θα υπάρχουν και σωστές προδιαγραφές θέλω να αναφερθώ στην προστασία του καταναλωτή. Όσο περισσότερο κοιτώ το θέμα αυτό, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνουμε ότι πρέπει να πάρουμε το θέμα αυτό πιο σοβαρά, διότι μέχρι το 2010 ε, τα τρία τέταρτα του διαθεσίμου εισοδήματος των δυτικοευρωπαϊκών ε, θα καλύπτεται σε άτομα που είναι πάνω από 50 ετών. Και τότε ε, έχουμε διάφορα προβλήματα σχετικά με την προστασία του καταναλωτικού για τον γυράσκοντα πληθυσμό, τις δημογραφικά προβλήματα και τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε επίσης και αυτό με οδηγεί στο θέμα της ψηφιακής οικονομίας και της ψηφιακής εποχής. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να μείνουν πίσω. Χρειάζεται ποιότητα για όλους τους καταναλωτές. Ε, σας ευχαριστώ, θα μας λείψετε και σας εύχομαι ε, κάθε επιτυχία στην επόμενη Γενική Διεύθυνση που θα αναλάβετε. Ευχαριστώ. Έχω προσθήσει τώρα και άλλους ομιλητές, ελπίζω να είστε πολύ σύντομοι, αλλά δεν θέλω καμία ομάδα να μείνει χωρίς φωνή. Κλείνω τώρα τον κατάλογο των ομιλητών στον κύριο Σαλβίνη για να μπορέσουμε γύρω στις 10 και 4 να έχουμε ολοκληρώσει και δίνω το λόγο στην ε, αντιπρόεδρό μου η οποία εργάζεται σκληρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη διότι η ώρα περνάει. Και όπως όλοι οι άλλοι θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο. Νομίζω ότι δουλέψαν πολύ σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω διότι ακόμη και αν δεν συμφωνούμε πάντοτε όπως είπε η κυρία Γκέπχαρτ η ειλικρίνειά σας και η συνεργασία σας σε όλες τις προτάσεις μας μας ικανοποίησε πολύ και ελπίζω ότι το ίδιο θα συμβεί και με τον αντικαταστάτη σας. Ε, θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον αντικαταστάτη σας διότι είσαστε υπεύθυνοι για τη μεταβατική περίοδο. Μιλήσατε για την ασφάλεια των προϊόντων και την ευελιξία των ε, επιγόντων μέτρων διότι πρέπει να δούμε πώς ε, αντιδρούν τα επίγοντα μέτρα για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων για να καταπολεμήσουμε μία φοβερή πληγή που είναι η παραποίηση, τα, ε, τα ε, αντίγραφα τα οποία αγοράζει κανείς στο ίντερνετ ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο μέλλον θα πρέπει ε, να υπάρξει μία σήμανση η οποία θα είναι πολύ ακριβής ε, να μπορούμε να ελέγχουμε τα προϊόντα και μάλιστα ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει ε, μεγάλης παρακολουθήσεως. Σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ συνάδελφοι να είστε ήσυχοι. Εάν θέλετε να συζητήσετε εκτός της οθούσης παρακαλώ για να ακούει κανείς τι έχετε να πείτε. Κυρία Μπίλτς, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Κούνεβα όπως και προλαλήσαντε για την προσήλωσή της, για τη φρεσκάδα της, διότι βλέπω ότι σας αρέσει να ε, δείχνετε ότι μία γυναίκα μπορεί να συμβάλλει στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Και ευχαριστώ και για την ε, πολιτική σας διαθήκη, ε, για την συνεννόηση και τη συνένεση στο Κοινοβούλιο, που είναι πολύ σημαντικό για αυτή την Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι διάβαζα το blog σας πριν γίνω και Ευρωβουλευτήνα και το εκτιμούσα πολύ, με βοήθησε πολύ και σας εύχομαι κάθε καλή επιτυχία για το μέλλον. Ευχαριστώ. Μπορείτε να συνεχίσετε το blog και να μας λέτε τι γίνεται, να μας δίνετε συμβουλές μέσω του blog. Ο κύριος Κόζουτσεκ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι εν ονόματι του ΕΛΚ θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο Κούνεβα για την συνεργασία της, για την προσήλωσή της. Είμαστε νέοι, αλλά η κυρία Κουνέβα αμέσως μας ε, προθυμοποιήθηκε να συνεργαστεί μαζί μας για την πρόοδο της εσωτερικής αγοράς και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Οι, πιο εύγλωτες είναι οι σύντομες παρεμβάσεις. Η κυρία Τούν. Ευχαριστώ. Η συνάδελφός μας η κυρία Γκέπχαρτ είπε ότι εργαζόμαστε για τους ανθρώπους και όχι για την εσωτερική αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι ε, αυτό ήταν η δύναμή σας κυρία Επίτροπε. Ε, φέρατε πολύ κοντά στον πολίτη το μήνυμα ότι η εσωτερική αγορά είναι προς όφελός του και ε, αναφερθήκατε σε διάφορα επιχειρήματα, δηλαδή ε, οι πολίτες στα κράτη-μέλη κατάλαβαν πόσο σημαντική είναι η λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς και μέσω της σωστής λειτουργίας εσωτερικής αγοράς. Αυτό το μήνυμα, η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά, οι προκλήσεις της εσωτερικής αγοράς είναι ένα μήνυμα το οποίο φέρατε κοντά στον πολίτη και βλέπω εδώ το μέλη της ομάδας σας που συμμετείχαν σε αυτές τις δράσεις τις ενημερωτικές. Θα συνεχίσουμε στην Επιτροπή μας και θα οργανώνουμε ε, συνεδριάσεις και ε, ε, συνέδρια και ελπίζουμε το μήνυμά σας θα περάσει σε όλους τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίοι θα εργαστούν σαν πρεσβευτές για την προώθηση των ε, επιτευγμάτων σας και για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς που πρέπει να πλησιάσει τους πολίτες για να μπορούν οι πολίτες να λειτουργούν καλύτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω. Τέλος ο κύριος Σαβίνη. Σας ευχαριστώ. Και εξ ονόματο ε, της ομάδας Ευρώπη τη Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Σα ευχαριστώ για την εργασία σα μέχρι τώρα μέχρι στιγμής ε, ε, συμφωνήσαμε και ακούσαμε και το αίτημα παρέμβαση όχι μόνο για τις εισαγωγές και την κατασκευή ε, προϊόντων κοντρεφασών αλλά και για την συναρμολόγησή τους γιατί είχαμε επαφέ με παραγωγούς ε, ρολογοπίες, ε, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία ε, και Ηνωμένο Βασίλειο και από ό,τι φαίνεται δεν φτάνει πλέον το ρολόι μαϊμού, αλλά τα διάφορα ανταλλακτικά του και κατασκευάζεται μετά εδώ, στην Ευρώπη. Οπότε πέραν αυτή τη υπόθεση ε, βρίσκονται αφοπλισμένε οι εταιρείε ε, που τα κατασκευάζουν. Πραγματικά το eBay και το ίντερνετ, ε, μάλιστα είχαμε μια υπόθεση που κέρδισε ο Λουί Βοητών κατά το eBay γιατί εκεί πολλούνταν προϊόντα κοντρεφασών. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τη δουλειά σας μέχρι στιγμής. Θα πρέπει να προσέξουμε και για όλα αυτά τα προϊόντα που είναι απομιμήσεις. Επίτροπε, πολλά αναφέρθηκαν, πολλά σημεία εθίχθησαν και θα ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε και να πάρετε και για τελευταία φορά το λόγο, αφού είναι η τελευταία φορά που θα είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μου χαρά και τιμή να ακούσω τις ε, σκέψεις για την πολιτική καταναλωτή. Και συμφωνώ με πολλά από όσα υπόθηκαν. Νομίζω πως ε, ζούμε σε πολύ ε, ενδιαφέροντες καιρούς. Θα μπορούσε να υπάρξει μια βελτίωση μέσω της πολύτιμης συνεισφοράς σας Ορισμένες σκέψεις είναι πιο πολιτικής φύσης. Η πρώτη αφορά τις αγορές και συμφωνώ με όσους λένε ότι πρόκειται για μια τόσο σημαντική υπόθεση. Όχι μόνο οι αγορές πρέπει να δουλεύουν για τον κόσμο, αλλά πρέπει να δουλεύουν για την ανάκτηση, για τις ε, θέσεις απασχόλησης και για την παγκόσμια επιτυχία. Νομίζω πως η πολιτική καταναλωτή δεν είναι απλά η πολιτική για τους καταναλωτές, αλλά είναι και η πολιτική για την αγορά. Και για τις επιχειρήσεις που είναι επίσης υπεύθυνε. Να πω κάτι ακόμα μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής καταναλωτή και αυτό είναι η, Ευρώπη, η ατζέντα Ευρώπη 2020. Θα ακούτε όλο ένα και περισσότερα πράγματα από την Κομισιόν για αυτή την στρατηγική και από τον Πρόεδρο Βαρόζο, αλλά θα ήθελα να σας πω ότι σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, οι υγιείς αγορές που ενημερώνουν τους καταναλωτές θα δημιουργήσουν πωλήσει, θέσεις απασχόλησης και θα αποφέρουν ε, κέρδη. Αυτές είναι οι ιδέες ε, τις οποίες, και μια σταθερά την οποία θα ακολουθήσει η Κομισιόν. Φυσικά και δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας όσον αφορά την ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα σε μια περίοδο ύφεση. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειε, αλλά ε, όταν περικόπτουμε τι δημόσιε δαπάνε, χρειάζεται ακόμα περισσότερο να δώσουμε και να προωθήσουμε τους καταναλωτές και να τους ενημερώσουμε γιατί θα μπορούσαν να κάνουν μια επιπλέον εργασία από την άποψη του κοινού του δημοσίου συμφέροντος. Κάποιες σκέψεις για τα όσα είπε ο κύριος Σβάμπ για τη συνεργασία. Εγώ αναγνωρίζω την σημασία της συνεργασίας. Για το θέμα της κυρίας Γκέπχαρτ πιστεύω πως ανέκαθεν λέγαμε πως η αποστολή μας είναι να φτιάξουμε μια εσωτερική αγορά που προσφέρει στους καταναλωτές όσον αφορά τις επιλογές ασφάλειας, και είπα και σαφώς ότι όλα τα προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να είναι ασφαλή, άσχετα από οποιαδήποτε συμ... σήμανση. Η ασφάλεια δεν είναι εθελοντική ή προαιρετική. Αυτή την ε, γραμμή θα πρέπει νομίζω να την ακολουθήσουμε. Για την παρατήρηση του κυρίου Γκρότσμαρκ, ε, ναι, έχετε δίκιο. Η εσωτερική αγορά ενισχύει τις ε, κανόνες για την ανιχνεσιμότητα και η εποπτεία της αγοράς, όπως είπα, και εδώ συμφωνούμε 100%, θα πρέπει να αναπτυχθεί με βάση δύο δυνάμεις τη Ένωση και αναφέρατε την αλληλεγγύη που είναι ένα πολύ κρίσιμο τομέα επιτυχία παγκοσμίω και αυτός ήταν, ε, αυτή ήταν μια από τι προτεραιότητε τη δικές μου δράση, Συμφωνώ μαζί σα, ότι αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στα επόμενα χρόνια. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα, ε, αλλά ε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για αυτή την ιδέα για το ερώτημα του κυρίου Τρενταφυλλίδη. Θα διατηρήσουμε την προσοχή μας στην παγκόσμια λυσίδα παραγωγής, γιατί οι καταναλωτές πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη ότι δεν γίνονται υποχωρήσεις όσον αφορά την ασφάλεια, τόσο για τα παιχνίδια όσο και για τα χριστουγεννιώτικα φώτα. Στην, στην παγκόσμια οικονομία η παγκόσμια ασφάλεια είναι ε, ένα αγαθό. Μαζί με τα κράτα-μέλη μας και την ε, αρχή παγκόσμια υποπτήρας, η Ευρώπη θα συνεχίσει να διασφαλίζει πως δεν θα υπάρχουν ε, κενά στην παγκόσμια παραγωγή. Οι ενεργοί δραστήριοι καταναλωτές είναι πολύ σημαντικοί στην παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας μαζί μου. Για την κυρία τη Σάλτερ Μόζε να πω ότι οι κυβερνήσεις ναι, θα πρέπει να αφιερώσουν περισσότερους πόρους για την εποπτεία της αγοράς. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ιδρυτικοί πατέρες της Ευρώπης επέλεξαν να έχουν ανοιχτή αγορά στην ε, Ευρώπη και η πραγματική εποπτεία της αγοράς είναι ένας πυλώνας για αυτήν την ε, επιλογή, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε καταφέρει να δώσουμε στον κόσμο την ε, ασφάλεια που είναι απαραίτητη. Για την ερώτηση της κυρίας Βάιλερ για τα χριστουγεννιάτικα φώτα. Σήμερα παρουσιάζουμε την κοινή δράση ε, των αρχών εποπτείας κρατών μελών. Αυτή η δράση έχει συνεχιστεί εδώ και κάποιους μήνες και έχει επιφέρει δύο θετικά αποτελέσματα. Πρώτον, η δοκιμή και η απόσυρση πολλών επικινδύνων προϊόντων και η συνειδητοποίηση και ενημέρωση για επιχειρήσεις, ε, καταναλωτές και αρχές καταναλωτή για αυτό το θέμα. Θα μπορούσα να σας δώσω το έγγραφο και να μιλήσουμε πιο εκτεταμένα για το θέμα. Για την ερώτηση της κυρία Στήλερ για τα μη ασφαλή σολάριουμ ή όροι οι προϋποθέσεις ασφάλειας δεν απαιτούν ε, όριο για την ε, ραδιενέργεια υπέρυθρων ε, ακτινών σε αυτά τα σε, αυτά τα σολάρια μου. και είμαι βέβαιη ότι οι κανόνες αυτοί όταν επιβάλλονται σωστά αρκούν για να προστατεύσουν τους καταναλωτές. Δεν θέλω εγώ να αντιγράφω κάθε απαγόρευση που ακούω ε, να επιβάλλεται σε άλλα μέρη του κόσμου αν αυτό σημαίνει την ε, περιορισμό της επιλογής του καταναλωτή. Δεν είναι αυτή η προσέγγιση μας. Εγώ συναντήθηκα με εκπροσώπους της ε, βιομηχανίας κατασκευής των Solarium για να συζητήσουμε το θέμα. Θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τον επόμενο χρόνο κοινέ δράσεις για αυτόν τον τομέα για την κυρία Μπερναντέτ Βερνιό, επειδή η επιβολή είναι πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, αναγνωρίζω απόλυτα αυτές τις προκλήσεις και όπω και ο Πρόεδρο Μπαρόζο πρόσφατα τόνισε, η επιβολή παραμένει πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει πολλά δικαιώματα καινούργια στου πολίτες της, αλλά ακόμα πρέπει να περάσει πολύ καιρό μέχρι ότου αυτά τα δικαιώματα να μετατραπούν σε πραγματικότητα. Γι' αυτό και η Κομισιόν έχει κάνει μια ανακοίνωση που στόχο έχει να καταστήσει την επιβολή πιο αποτελεσματική και συνεπή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν γέννη, ναι, θα, για το blog θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Ελπίζω πως θα χρησιμοποιήσετε με περισσότερο πολιτικό τρόπο το δίκτυο όχι μόνο για να παίρνετε τα πρακτικά, αλλά για να υπάρξει μια δημοκρατία μέσω ίντερνετ. Ίσως ήταν ένα επόμενο βήμα. Είναι πραγματικά ένας ε, μελλοντικός καινούριος κόσμος που μας περιμένει. Για τα ευγενικά λόγια του κύριου Κόσμη και σας ευχαριστώ. Η προστασία του καταναλωτή είναι στην κορυφή της πολιτικής ατζέντα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα προϊόντα και τις σχετικές πολιτικές και είμαι βέβαιος πως η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο θα συνεχίσουν να εργάζονται από αυτόν. Για την κυρία Τούν, στόχος μου ήταν να Έχουμε την εσωτερική αγορά στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών. Για Ευρώπη, για όλους. Για τον κύριο Σαφίνη, οι απομιμήσεις πραγματικά είναι μία πρόκληση και μία κατάρα για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για τα την πολιτική καταναλωτή, ωστόσο μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση υποπτήρια τη αγοράς που θα καλύπτει τις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και προπαροχής είναι πολύ κρίσιμη για την επιτυχία στον απογόνα κατά των απομιμήσεων. Το ίδιο είναι και η εκπαίδευση των καταναλωτών. Να πούμε στους καταναλωτές ότι τον αγοράζουν απομιμήσεις δεν είναι ε, κάτι το οποίο είναι ε, καλό. Κοστίζει ευρωπαϊκές θέσεις και Θυμάμαι την πρώτη μου συμμετοχή εδώ, ήταν ε, πριν την ακρόαση και σας είπα ότι θα ήθελα να δω την αγορά ως έναν τον άνθρωπο του Νταβίντσι. Και, ελπίζω πως αυτό, ε, και νομίζω πως αυτό θα παραμείνει έργο για τα επόμενα χρόνια. Το να δεχτούμε το status quo σημαίνει ότι πάμε πίσω, ότι υποχωρούμε, οπισθοχωρούμε. Είστε εξαιρετικοί εταίροι, ωστόσο μπορεί να, συμφωνώ, να διαφωνούμε. Είναι υγιής η διαφωνία αυτή και είμαι βέβαιος πως ε, τα κοινά στοιχεία είναι τα περισσότερα και εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Uh, well, uh, Commissioner, um, I think the war... Επίτροπε, νομίζω πως... Ε, η θερμότητα με την οποία σας υποδεχθήκαμε και ο χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις ε, των συναδέλφων από μόνα τους μιλούν για την συνεργασία μας. Ε, το είδαμε εξ αρχής στην τελευταία θητεία που ήρθατε εδώ το Φεβρουάριο του 2007 ήταν η πρώτη πιθανή ευκαιρία και ήδη έχετε πολλούς φίλους και έχετε νομίζω εντυπωσιάσει και τους συναδέλφους που μόλις ήρθαν τον περασμένο Ιούνιο. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον. Νομίζω πως μεγάλη ευθύνη έχει αυτή η Επιτροπή. Μιλήσαμε με την κυρία Γκέπχαρτ και ο κύριος Βάπ το ανέφερε τα θέματα και τις ανησυχίες μας για τον μελλοντικό συντονισμό των δραστηριότητων με τη νέα Επιτροπή και εγώ θα στείλω επιστολή στον πρόεδρο Μπαρόζο. Οι συντονιστές με μου ζήτησαν να το κάνω, αλλά νομίζω πως ε, αυτός ο συντονισμός ε, είναι απαραίτητο. Κοιτάμε διάφορου παράγοντε. Μπορεί να επεκταθούμε και στα τελωνία, όπω αναφέρατε, ένα άλλο τομέα συντονισμού. Νομίζω μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι οι συνάδελφοι και η Επιτροπή μας ε, θα αναλάβουν αυτή την ευθύνη πολύ σοβαρά. μπορείτε να δώσετε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Μας δώσετε ένα ισχυρό μήνυμα και εμείς ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τις επόμενες προκλήσεις που μπορεί να αναλάβετε. Ίσως ήταν μεγάλη πρωταθλήτρια ε, υπέρ των καταναλωτών της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε. Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή να συνεργαστούμε μαζί σας. Ε, Äh, Πρόεδρε, έχει επαναληφθεί ένα πρόβλημα για το οποίο λυπούμε πάρα πολύ. Η συνάδελφός μου Ζωζέφ Άντρες Μπαρέα ξαναέφυγε διότι δεν υπήρχε μετάφραση προς Ισπανικά και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να συμμετάσχει στην ε, συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, δεν μπορεί ε, να ε, διαιωνίζεται, το έχω επισημάνει επανειλημμένος και δεν είναι δυνατόν να μην έχουν οι διερμηνείς γλώσσες οι οποίες είναι δικές τους για να ακούν και να μπορούν να μιλήσουν. Ναι, όπως ξέρετε όμως ε, ε, αυτή η Επιτροπή έχει συνήθως λίγες γλώσσες. Ε, για μένα είναι βασική ημέρα αυτή. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μία ψηφοφορία. Ελπίζω να συνεργαστείτε μαζί μου. Θα, όπως είχα πει, οι ψηφοφορίες θα γίνουν με το χέρι και όχι με ηλεκτρονικές κάρτες ε, και θα πρέπει να ξέρω που κάθε ο καθένας. Είναι όμως η πρώτη φορά και καλό θα ήταν να ελέγξουμε ποιος πρόκειται να ψηφίσει για ποια ομάδα. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο να, ε, μιλήσω, να δούμε ποιοι είναι εδώ από τους υπευθύνους της Επιτροπής και θα ήθελα να παρακαλέσω όσους ε, ψηφίζουν να μου πούν. Το ΕΛΚ έχει 14 ψήφους. Μπορώ να ζητήσω λοιπόν ε, από το ΕΛΚ να μας πούν ποιοι είναι. Έχουμε τους 14. Μπορούμε να ελέγξουμε μήπως έχουμε περισσότερους από 14. Ναι, και ο κύριος Είναι βασικό να ξέρουμε ποιος είναι στην πίσω μεριά. Μετά, οι σοσιαλιστές έχουν δέκα. Μπορώ να παρακαλέσω τους σοσιαλιστές να, μας, να σηκώσουν το χέρι τους. Οι φιλελεύθεροι έχουν τέσσερις. Ο κύριος Μπεζόη δεν με ακούει, αλλά μ' άκουσε τώρα. Οι πράσινοι έχουν τρεις. Οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί έχουν τρεις. Εγώ δεν θα ψηφίζω εάν είσαστε τρεις εκεί. Ούτως ή άλλως έχω αρκετά να κάνω, δεν χρειάζεται να ψηφίζω κιόλας. Ε, δύο ε, δύο γκουε, δύο EFD. Εντάξει, ευχαριστώ. Η πρώτη ψηφοφορία είναι για τον πίνακα αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή ήταν η πρώτη μου έκθεση, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για καλή συνεργασία μαζί σας, ιδίω με τους Σκιώδης και την ε, Γραμματεία, η Μίνα Πετρούτσι και σας ευχαριστώ πολύ Είχα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευρεία στήριξη, διότι πολλοί είπαν ότι υπάρχει μία νέα πνοή ε, και κίνηση στην εσωτερική αγορά. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένη, διότι μετά από τόσες συνεδριάσεις που είχαμε χθες το βράδυ ή την τελευταία στιγμή, απροσδόκητα έρχεται η φωνή των συναδέλφων σοσιαλιστών που απορρίπτουν μία τροπολογία που είναι σημαντική σχετικά με τη δοκιμασία της εσωτερικής αγοράς. Και νομίζω ότι είναι μια επίδειξη δυνάμεως σε αυτή την Επιτροπή. και προσπαθούν να επηρεάζουν την την επίδραση του εγγράφου αυτού στην εσωτερική αγορά. Ελπίζω όμως ότι θα έχουμε θετικές ε, ε, ε, θετική έκβαση. Σας χαιρετίζω την αθρώα παρουσίαση σήμερα στην ψηφοφορία. Ε, δεν θέλω να ε, ξεκινήσω μια ευρία συζήτηση από αυτό, αλλά βλέπω ο κύριος Βόμουνα που ζητάει το λόγο. Ε, βλέπω ότι έχουμε ένα κείμενο πολύ επικοδομητικό. Δυστυχώς η τροπολογία 19 που θα μπορούσε να οδηγήσει σε, μία, σε ένα συμβιβασμό είναι πολύ δογματική θα μπορούσατε να την έχετε αποσύρει και δυστυχώς ε, ε, έχουμε μία ε, αρνητική έκβαση σε εργασίες οι οποίες γενικά είχαν διεξαχθεί σε καλό πνεύμα και την τροπολογία αυτή θα την καταψηφίσουμε. Λοιπόν, παράγραφος 2, τροπολογία 8, ποιος είναι υπέρ. Carried by a large majority. Ε, εγκρίνεται με μεγάλη ψήφο ε, ε, η τροπολογία του κυρίου Νόκ υπέρ κατά τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Οπότε οι τροπολογίες 9 και 10 ε, καταπίπτουν. Ε, τροπολογία που πάει εκεί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Ε, ποιος είναι υπέρ. Those against. That was, was 15 in favor. 15 υπέρ, 21 κατά, άρα κατεψηφίσει. Τώρα στην τροπολογία 14 έχουμε μία α, προφορική τροπολογία της κυρίας Λούκεγκάρντ, οπότε α, ε, θα την ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Two against. That's carried. Κατά uh, amendment Καταπίπτει ε, η, τροπολογία, ε, ε, η τροπολογία 15 υπέρ. Κατά εγκρίνεται η τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 15 υπέρ, 22 κατά. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ αυτής της συμβασικής τροπολογίας. Κατά. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα θα περάσουμε στην παράγραφο 6. Ε, τροπολογία υπέρ, 19 υπέρ 22 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 22 υπέρ και 15 κατά. Η 20 έχει αποσυρθεί. 21 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται ομόφωνα. Παράγραφος 6 νέα. Και πάλι προφορική τροπολογία. Ο κ. Λόκαγκαρτ την εγκρίνει. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. εγκρίνεται 25 υπέρ 12 κατά. Η, τροπολογία, η αρχική τροπολογία 22 καταπίπτει. Παράγραφος 7α. Υπάρχει πάλι μια προφορική τροπολογία ε, τροπολογία 23. Ε, ε, ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ εγκρίνεται ομόφωνα. Τώρα θα περάσουμε στην παράγραφο 9, γιατί 24 έχει αποσυρθεί και 25 έχει αποσυρθεί. Ε, παράγραφος 10, τροπολογία 26, υπέρ. Ψηφικατά, όχι, εγκρίνεται ομόφωνα. Η 27 έχει αποσυρθεί, η 28 έχει αποσυρθεί και θα περάσουμε στην 29. Υπέρ παρακαλώ. Υπάρχουν ψηφικατά. Δύο κατά, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα, συμβιβαστική ε, τροπολογία 3 για την παράγραφο 12, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται ομόφωνα. Ε, οι τροπολογίες 30-31 καταπίπτουν και θα περάσουμε στη 32. Ε, στην παράγραφο 13, υπέρ παρακαλώ. Κατά, εγκρίνεται. Η 33, υπέρ κατά εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Η 34 τώρα, υπέρ παρακαλώ. Κατά και πάλι εγκρίνεται με σημαντική πλειοψηφία. 35 υπέρ. Υπάρχουν ψήφοι κατά. Όχι, εγκρίνεται ομόφωνα. 36 υπέρ. Κατά, εγκρίνεται και πάλι ομόφωνα. Τώρα είμαστε σε ιδεολογικές σκέψεις. Έχουμε μια προφορική τροπολογία σε προφορική σκέψη μόνο 1. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται ομόφωνα. Η αρχική λοιπόν τροπολογία καταπίπτει. Ε, τροπολογία 2 στο G. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία παριθμών 3 στο H, στο Ι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με πλειοψηφία το 4 στο M. MA, νέο, υπέρ. Υπάρχουν ψηφικατά. Όχι, εγκρίνεται ομόφωνα. Ετολογική σκέψη O. Ετροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Ομόφωνα εγκρίνεται. OA ο α, α. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται ομόφωνα. Ε, τροπολογία 7. Υπέρ, κατά. Και τώρα θα έρθουμε στην τελική ψηφοφορία, ολόκληρη την έκθεση. Ποιος είναι υπέρ του τελικού κειμένου. Υπέρ. Those against. Κατά. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 15 κατά. So like to... Ωραία λοιπόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τούν και να τη συγχαρώ για την ολοκλήρωση της πρώτης της έκθεσης. Ε, βεβαίως ε, θα πάει στην Ολομέλεια. Βεβαίως θα θέλαμε να έχουμε μια σύντηση μεταξύ των ομάδων για να δούμε κατά πόσο υπάρχει μια πλήρης υποστήριξη στην Ολομέλεια. Τώρα θα περάσουμε στην επόμενη έκθεση για τον ε, εφοδιασμό με φυσικό αέριο της κυρίας Κανιέτε. Και της κυρία Κανιέτε είναι η πρώτη της έκθεση. Ε, συγχαρητήρια κυρία Κανιέτε. Ε, κύριε Χάνσεν, θέλετε να πείτε κάτι. Bardzo przepraszam, że przed panią sprawozdawcą e, zabieram głos, ale e, zostałam zobowiązana przez pana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 Uh, Article 1, Amendment 30. Those in favour? Those against? Carried. Υπέρ παρακαλώ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, που έχει ψηφιστεί σαν μια προσθήκη στο άρθρο 1. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται με μεγάλη ψηφιφυρία. Ε, ε, πλειοψηφία, συγγνώμη. Η 2 έχει αποσυρθεί. Έχουμε μια συμβεστική τροπολογία από τρεις πολιτικές ομάδες. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται και στη συνέχεια... Οι 32, 33, 34 καταπίπτουν και 35 περνάμε στην 36. Ποιοι είναι υπέρ της 36, κατά, απορρίπτεται. Και τώρα θα περάσουμε στο άρθρο 3, τροπολογία 37. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται ομόφωνα. Τροπολογία 4 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με μεγάλη ε, πλειοψηφία. 39. Υπέρ κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 40, υπέρ, κατά, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 41, υπέρ, κατά, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 40, η 42 έχει αποσυρθεί, 43 τώρα, υπέρ, κατά, απορρίπτεται η προφορική τροπολογία του κ. Μάντερς 44. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται ομόφωνα. Η τροπολογία 44 καταπίπτει και τώρα θα περάσουμε στη 47 που είναι και πάλι μια προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά εγκρίνεται ομόφωνα. Τώρα θα περάσουμε στη συμβαστική τροπολογία 2 από τέτοιες πολιτικές ομάδες υπέρ της συμβαστικη τροπολογίας. Κατά εγκρίνεται ομόφωνα. 48 και 49 περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 3 εκ μέρους των πολιτικών ομάδων υπέρ της συμβαστική τροπολογίας 3. Κατά εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία. Οι 51 και 52 καταπίπτουν, οι 53, 54, 55 έχουν αποσυρθεί, έτσι περνάμε στην 6 της εισηγήτριας για το άρθρο 9, υπέρ. Κατά, εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία. Οι 56 έχουν αποσυρθεί. Οι 57 τώρα, υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. Άρθρο 10. Συμβαστική ερωπολογία 4 εκ μέρους τεσσάρων πολιτικών ομάδων. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται ομόφωνα. Όχι, υπάρχουν τρεις αποχές. Ωραία, με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Οι 59 και 58 καταπίπτουν και περνάμε στην 60. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Η 61 έχει αποσυρθεί. 62 υπέρ. Υπέρ της 62. Πολλοί συνάδελφοι και η κυρία Χάνσλικ.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 13. 13, 14, 15, 17, 18, 14. 14, 15, 16. Yeah. 16. 16. Okay, so that's carried. Ωραία, λοιπόν, εγκρίνεται 19 προς 16. Τώρα θα περάσουμε στο άρθρο 11, τροπολογία 63 του Τουάν Μάντερς, υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. Άρθρο 12. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται μεγάλη πλειοψηφία. 66 και 67 έχουν αποσυρθεί και τώρα είμαστε στην αιτιολογική σκέψη 4 με μία προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7. Υπέρ κατά εγκρίνεται ομόφωνα. Στη συνέχεια περνάμε στην τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ετυλογική σκέψη 6. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Όχι, εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος. Οι τροπολογίες 11 και 12 έχουν αποσυρθεί. Η τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. απορρίπτεται. Η τροπολογία 14 στην λογική σκέψη 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά απορρίπτεται. Η 16 στην σκέψη 13 υπέρ κατά εγκρίνεται. Η 17 στην σκέψη 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τελική σκέψη 15. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 17 έχει αποσυρθεί. Και τώρα θα περάσουμε στη συμβαστική τροπολογία 5, Συνολική σκέψη 18. Υπέρ. Υπάρχουν ψήφοι κατά. Και τρεις αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν με τρεις αποχές. Οι 21, 23, 24 και 25 καταπίπτουν και θα περάσουμε στην 26 με μια προφορική τροπολογία του Τόεν Μάντερς. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στην δηλογική σκέψη 21. Έχει αποσυρθεί 27. Είμαι στην δηλογική σκέψη 23. Η τροπολογία 28 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 29 στην αιτιολογική σκέψη 29. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα θα έρθουμε στην τελική ψηφοφορία. Υπέρ. Uh, κατά. Δύο κατά. Εγκρίνεται λοιπόν με πλατιά πλειοψηφία, δύο ψήφοι κατά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κανιέτε Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή είναι μια γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής. Θα πρέπει λοιπόν να επρασπίσουμε την άποψή μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, στην Επιτροπή Βιομηχανίας, λέει ο Πρόεδρος. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που συμμετείχατε στη ψηφοφορία σήμερα το πρωί και θα σας δώσω λίγα λεπτά να καθίσετε και θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Okay, we have got other business, so could I ask you please... Έχουμε και, άλλες, και άλλα θέματα, οπότε παρακαλώ όσοι θέλετε να φύγετε, να φύγετε ησύχω, ώστε να προχωρήσουμε. Γιατί έχουμε ένα έγγραφο για τον προπολογισμό να εξετάσουμε. Uh, so, um, could you please carry on conversations outside the room, please, uh, so we can have a bit of quiet for our rapporteur. So now we're going to... Um... Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσουμε και θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης που θα πάει στην Επιτροπή Ελέγχου, Πληροφο... Ελέγχου Προπολογισμού για την απαλλαγή του Γενικού Προπολογισμού για το οικονομικό έτος για τις πτυχές που αφορούν τη δική μας επιτροπή. Έχουμε εδώ τον εισηγητή κύριο Λίμαν και για τους σκιώδες, τον κύριο Γκρέχα, Λιρόι. Λοιπόν, κύριε μου θέλετε να παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Να ευχαριστώ. Για μένα είναι η πρώτη μου έκθεση πρώτο σχέδιο έκθεσης, γνωμοδότησης μάλλον. Και μπορώ να σας πω ότι είναι πολύ ωραία η εμπειρία. Παρακαλώ ησυχία. Όπως σας είπα, είναι καλή εμπειρία να δουλέψουμε, με, συνεργαστούμε με όλους τους ε, ε, συνεργάτες της Επιτροπής και από την πολιτική μας ομάδα για να συντάξουμε αυτήν την έκθεση. Ε, καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη γιατί κάποιες μεταφράσεις δεν είναι ακόμα έτοιμες. Δεν είναι δικό μου το σφάλμα. Έχουμε μόνο την αγγλική εκδοχή της γνωμοδότησης και περιμένουμε ακόμα το γερμανικό και γαλλικό κείμενο αλλά θα το έχετε πριν από τις 9 Δεκεμβρίου και όλοι οι μεταφραστές εργάζονται πολύ σκληρά για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Όπως είδατε, είναι μια σύντομη γνωμοδότηση που περιλαμβάνει πέντε παρατηρήσεις για το θέμα. Νομίζω πως και τα πέντε θέματα είναι σαφή. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ σε όλα όσα έχω γράψει. Απλώς θα επιστήσω την προσοχή σας στο σημείο 4 που αφορά το πρόγραμμα Solvit. Πολλά χρήματα το 2008 δεν χρησιμοποιήθηκαν, από ό,τι φαίνεται. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό το πρόγραμμα το 2008 και τα στοιχεία για το 2009 θα είναι πολύ καλύτερα. Πολλά από τα χρήματα ήδη έχουν ε, προγραμματιστεί για την δαπάνη τους. Δεν απορροφήθηκαν λοιπόν όλα τα χρήματα, αλλά σίγουρα για το 2009 τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Γι' αυτό ε, δεν έχω να κάνω πολλές παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, για την ώρα. Σας ευχαριστώ. εστιάζουμε σε κάποια σημεία κλειδιά. Θα δώσω το λόγο και στους σκιώδες Γιατί Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Γκρούμπεν και την κυρία Τεβέτ από την Γενική Διεύθυνση της Κομισιόν που είναι αρμόδια. Ο κύριος Γκρέχ πρώτα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή για όλα αυτά τα θέματα. Έχω μόνο μία παρατήρηση που απευθύνεται στην Κομισιόν και είναι η ίδια για το θέμα του Solvit. Νομίζω πως ε, αυτό το συγκεκριμένο απόθεμα είχε δημιουργηθεί στον προπολογισμό του 2008 για να χρηματοδοτήσει το Solvit. Μόνο 48 προγράμματα ε, υπήρξαν και θα ήθελα να, δούμε, να δει η Κομισιόν ε, τι συμβαίνει το 2009 με το ίδιο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Θα το συζητήσουμε. Νομίζω ο κ. Μπουζό κάνει την έκθεση για το Solvit. Αλλά έχετε και το λόγο για τον προπολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα συμπεράσματα ε, της νομοδότησης. Επίσης θέλω να καλωσορίσω το ποσοστό εκτέλεσης για την ε, γραμμή 12.02.01 καθώς και για τα ε, πολιτική ε, τελωνίων και για το πρόγραμμα καταναλωτών. Έχουμε και συζήτηση σήμερα για το Solvit. Αυτά όλα συνέβησαν για το 2008. Το 2009 τα πράγματα φαίνονται πολύ πολύ καλύτερα και με τις προτάσεις που κάναμε από κοινού το 2010 και τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ μεγάλη βελτίωση σε αυτό το τομέα δηλαδή στο ποσοστά εκτέλεσης. Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο σημείο 3 για τα τελωνία. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική πτυχή για τα όσα συζητάμε εδώ και θα πρέπει να προσέξουμε τα όσα μας είπε ο εισηγητής εδώ. Για τους ελέγχους τους επιτόπιους που κάνουν το κράτη μελή. Φορτικά υποστηρίζω τα όσα γράφονται εδώ και περιμένω να συζητήσουμε την περισσότερες λεπτομέρειες στο Σόλβιτ, στο επόμενο σημείο που έχουμε χωριστή συζήτηση μόνο για το Σόλβιτ. Κυρία Ρούλερ, Μπορώ να συμφωνήσω με τους προλαλήσεντες, βρίσκω ότι η έκθεση είναι καλή, ε, συζητάμε για τα τελωνία διότι παραπονούμαστε εδώ και χρόνια ότι τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν επαρκές προσωπικό αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ε, ότι ε, οι, οι αποδίδονται στην Ευρωπαϊκή Επιστροπή αλλά κάτι πρέπει να κάνουν και τα κράτη και εδώ συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει ή δεν έχει εφαρμοστεί καλά το πρόγραμμα ή ε, ε, δεν επαρκεί. Ευχαριστώ κυρία Γκέπχαρτ. Τώρα και μετά κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η έκθεση είναι πολύ καλή και τα αναφέρεται στα βασικά θέματα τα οποία παριθμίζονται. Σχετικά με το 4 θα ήθελα να πω και να συμφωνήσω με αυτά που είπαν ήδη διάφοροι προλαλήσαντες, δηλαδή λυπούμε ότι δεν θα είμαι μετά στο Meet, γιατί πρέπει να πάω και στην αντιπροσωπεία της ε, Κίνας γιατί και εκεί όπως ξέρετε μιλάμε για την ασφάλεια των προϊόντων Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό και ελπίζω ότι και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι γίνεται με τη χρηματοδότηση διότι για τον προπολογισμό του 2008 είχαμε εισάγει αυτή την γραμμή ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει μία ενημερωτική εκστρατεία. Δεν είναι θέμα της Επιτροπής, είναι των κρατών μελών βεβαίως, αλλά είχαμε διαπιστώσει ότι ελάχιστοι πολίτες γνώριζαν το Solvit και εγώ όταν ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώθηκα ότι υπάρχει καν το Solvit και αυτή η δραστηριότητα. Είναι μία προσπάθεια για τους πολίτες, γι' αυτό και ζητήσαμε να υπάρξει μια ενημερωτική εκστρατεία κατά τρόπον ώστε οι εμπλεκόμενοι να ξέρουν ότι υπάρχει εκεί μία υπηρεσία στην οποία μπορούν είτε οι ίδιοι είτε τα κράτη του να στραφούν. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχω καταλάβει ε, τι έχει γίνει με αυτήν την ε, εκστρατεία πληροφόρησης παρόλο που ταξιδεύω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέχω και στη Γερμανία αλλά ε, δεν έχω διαπιστώσει να υπάρχει μια εκστρατεία ενημέρωση των πολιτών που να τους ενημερώνει ότι κάτι υπάρχει. Γι' αυτό και το σημείο 4 κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαμε κάπως να το αναδιατυπώσουμε διότι έτσι που είναι εδώ είναι σωστό μεν αλλά μπορεί κανείς να ε, καταλήξει στη λανθασμένη στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται χρηματοδότηση, η οποία είναι απαραίτητη για να καταλήξουμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και ο κύριος Μπόης, θέλουμε να δούμε την, την ε, συχνότητα των ελέγχων ε, στα κρατημέλη μελη Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να φροντίσουμε να συνεχιστεί. Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αφού ακούσαμε προηγουμένως από τον Επίτροπο την εντυπωτικοποίηση των ελέγχων, ακόμα και για τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια είδαμε, ανακαλύψαμε ότι υπήρχε κοινό πρόβλημα. Για το Solvit θα το συζητήσουμε στο επόμενο θέμα. Πολύ ενδιαφέρον ε, ο χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης. Με εκπλήσει το 40% μόνο εκτέλεση. Θα συζητήσουμε Εισηγητής της έκθεση είναι ο κ. Βαν Κάμπ. Ζητώ συγγνώμη κύριε Κάμπ γιατί σας μπέρδεψα με τον κύριο Μπουζόη. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι όταν μιλάμε για απαλλαγή και όταν βλέπουμε χαμηλά ποσοστά εκτέλεση θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό για να λύσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βαντεκά. Πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μάριαν Γκρούμπερ, που είναι τακτική επισκέπτρια στην Επιτροπή μας, εκπρόσωπος της Επιτροπής, για θέματα φορολογικά. Ευχαριστώ κύριε Χάρμπερ. Εγώ θέλω απλώ να διευκρινίσω και να καθησυχάσω την Επιτροπή, γιατί καταρχήν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη γραμμή Solvit που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2008. Ωστόσο, επειδή δεν είχαμε χωριστή δημοσιονομική γραμμή για το 2009, Ήδη ήμασταν σε ένα κύκλο δαπανών που βασιζόταν στον γενικό προϋπολογισμό για τα θέματα εσωτερικής αγοράς. Άρα, 48% εκτέλεση για το Solvit ε, το 2008 δεν είναι η πλήρης εικόνα. Είχαμε 100% ε, ε, αναλογία, ποσοστό δέσμευσης μάλλον για αυτό το προπολογισμό. Βέβαια, οι συμβάσεις ακόμα συνάπτωταν, οι υπηρεσίες παραδόθηκαν το 2009, άρα λοιπόν τα τιμολόγια τα λάβαμε μόνο το 2009. Αν δείτε τώρα λοιπόν την πλήρη εικόνα, το ποσοστό εκτέλεσης είναι κοντά στο 100% γιατί οι πληρωμές έγιναν τόσο το 2008 όσο και το 2009. Για τον προπολογισμό 2009 που είναι 800.000 έχουμε παρόμοια κατάσταση. Το ποσοστό δέσμευσης και το ποσοστό εκτέλεσης θα φτάσουν κοντά στο 100%. Και πάλι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τον προπολογισμό και προσπαθούμε να το δαπανούμε σωστά. Σε σχέση με τις ερωτήσεις της κυρίας Γκέπχαρτ για το τι ακριβώς κάναμε με τα χρήματα, μπορούμε να σας δώσουμε μια γενική εικόνα των δαπανών, αλλά για να συνοψίσω, να σας πω ότι η μεγάλη πλειοψηφία αφορούσε την πρόθεση υλικό πρόθεσης, γιατί η στρατηγική που έχουμε υιοθετήσει για την πρόθεση του Solvit λειτουργεί με πολλαπλασιαστές. Έχουμε προωθήσει το Solvit, α πούμε, μέχρι το δικτύο επιχειρήσεων, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή, το Europe Direct, όλες τις υπηρεσίες που είναι κοντά στου πολίτες. Βέβαια, με 200.000 ευρώ δεν μπορείς να κάνεις και πολύ ευρεία εκστρατεία μία, μία διαφήμιση στην εφημερίδα θα είχαν ξανεμιστεί τα χρήματα. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη λύση με τους πολλαπλασιαστές της διαφήμισης. Πρέπει να γίνει πιο στοχοθετημένη η διαφήμιση, γιατί αν δεν φτάσουμε στο σωστό κρατήριο, τότε κινδυνεύουν τα κέντρα Solvit να πλημμυρίσουν με κόσμο που δεν είναι για εκείνα. Θα συνεχίσουμε με αυτή τη στρατηγική για το 2010 και τον προπολογισμό αλλά θα σας τα πω αυτά στο επόμενο σημείο. Σας ευχαριστούμε για αυτή την διευκρίνηση. Είμαι σίγουρη ότι ο κ. Βαντεκάμ θα σας μιλήσει για αυτά τα θέματα και ιδιαίτερος. Ο κ. Δεβέτς, ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Εγώ θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια στο σημείο 3 όπου όπου εκφράζεται ε, το παράπονο πως ε, η συχνότητα των ελέγχων επιτοπίως είναι πολύ χαμηλή. Ίσως όμως να έχετε κάπως μπερδευτεί γιατί οι έλεγχοι αυτοί γίνονται για λόγους ασφαλείας όταν εισάγονται αγαθά στα σύνορα. Ενώ όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων είναι περισσότερο ex post έλεγχοι εγγράφων. Ε, τούτου λεχθέντος, η στρατηγική για, για την εφαρμογή των ελέγχων αυτών ε, είναι στρατηγική την οποία, για την οποία είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη. Δεν είναι αρμοδιότητα κοινοτική. Ωστόσο, η Κομισιόν ε, πάντοτε προσπαθεί να χρησιμοποιεί την ανάλυση κινδύνου για να εστιάσει στους εμπόρους υψηλού κινδύνου ή στα φορτία υψηλού κινδύνου. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να διευκολύνει για την καλύτερη χρήση των ανθρωπίνων πόρων. Οπότε στόχος της Κομισιόν εδώ είναι να προσπαθήσει να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στους ελέγχους και τη διευκόλυνση των ελέγχων για τους αξιόπιστους εμπόρους. Ευχαριστώ. Κύριε Βαντεκάμπα, να σας δώσω το λόγο για να συνοψίσετε. Με βάση τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Και ίσως μπορείτε να μας πείτε και δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της έκθεσής σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους κοιόδης εισηγητές για τα σχόλιά τους και επίση την Κομισιόν. Πρότασή μου είναι να επεκτείνουμε λίγο το κείμενο του 4, της παραγράφου 4, όπως είπε η κυρία Κέπαρτ, γιατί είναι το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής μας, πάει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και κάποια από όλα αυτά θα χαθούν. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν να τα επεκτείνουμε λίγο το σημείο 4 για το τι συνέβη το 2008 και να δούμε τα αποτελέσματα μετά το 2009 και 2010. Ίσως θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε κάποιες παρατηρήσεις για τους ε, επιτόπιους ελέγχους ε, από τα τοπικά τελωνία. Γιατί για παράδειγμα στις κάτω χώρες τα πάντα που ε, μάλλον ό,τι πάει καλά προέρχεται από την εθνική κυβέρνηση και ό,τι πάει στραβά φταίει η Ευρώπη. Ίσως χάσουμε κάποιες λεπτομέρειες, μπορούμε και να επεκτείνουμε κάπως το κείμενο και θα ήθελα να ζητήσω από τη Γραμματεία να μου δώσει κάποιες ακόμα προτάσεις. Δυστυχώς είμαι νέος σε αυτό το θέμα του χρονοδιαγράμματος. Κύριε Μάλκομ, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ο πρόεδρος έχει πάντα τις πληροφορίες αυτές. Οι ε, κανονικά θα ήθελα οι εισηγητέ να τις έχουν πριν από μένα. Εν πάση περιπτώσει, πρώτα, πρόταση είναι η προθεσμία υποβολής κατά τα τροπολογιών να είναι 18 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Οι άλλες γλωσσικές εκδοχές, όπως είπατε, θα είναι διαθέσιμες, οπότε θα έχετε και το χρόνο γι' αυτό. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα υιοθετήσουμε στην Επιτροπή 25 και 26 Ιανουαρίου 2010 και αυτό ίσως εξαρτηθεί κάπως αν θα παρατείνουμε και για τις 27 Ιανουαρίου που θα γίνει μια, ίσως μια ειδική ολομέλεια για να επιβεβαιωθεί ο διορισμός των νέων επιτρόπων οπότε θα πρέπει να παρατείνουμε. Εν πάση περιπτώσει θα είναι μέσα στην ε, ε, συνεδρίαση Ιανουαρίου της Επιτροπής. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού θα υιοθετήσει στις 2 Μαρτίου την έκθεσή της και θα περάσει τον Απρίλιο από την Ολομέλεια. Εντάξει. Άρα λοιπόν μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου έχετε συνάδελφοι για να προετοιμάσετε τις τροπολογίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βάντεκαμ που δούλεψε τόσο σκληρά στην πρώτη σας έκθεση. Ήσασταν πολύ μεθοδικός. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή και θα περιμένουμε το τελικό σας κείμενο. Τώρα θα περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σχέδιο έκθεσης που <laughs> πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας για το Solvit ε, ο κύριος Μπουσό είναι ο εισηγητής μας και θα ήθελα να τον καλωσορίσω. Οι εισηγητές, ε, οι σκιώδεις εισηγήτρες, συγγνώμη κυρία Ρόιτεβα, δεν την βλέπω εδώ. Και η κυρία Στάιλερ, η κυρία Ρούλερ, ο κύριος Σκόσκι, ο κύριος Ντέγιονγκ δεν είναι εδώ και ο κύριος Σαβίνη δεν είναι εδώ. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο. Η κυρία Γκρούμπε θα απαντήσει εκ μέρους της Επιτροπής. Δεν ξέρω, είναι εκεί πίσω. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μπουσόη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, διακριμένοι συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη που δεν ήμουν ε, εδώ σήμερα το πρωί, ήμουν στην Επιτροπή Προπολογισμών όπου έλαβε χώρα μια σημαντική ψηφοφορία και έχασα την ευκαιρία να πω στην ε, Επίτροπο κυρία Κούνεβη πόσο σημαντική ήταν η συνεργασία μας και πόσο σημαντική για την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση το Solvit θα έχει να δαπανίσει του χρόνου ένα εκατομμύριο. Με ενθαρρύνουν πάρα πολύ τα όσα υπόθηκαν, ότι μέχρι στιγμής όλα τα χρήματα έχουν αξιοποιηθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά. Τώρα, το σχέδιο πρότασης είναι ταυτόχρονα μία αξιολόγηση του προγράμματος Solvit και της αποτελεσματικότητάς του και ταυτόχρονα μία προσπάθεια βελτίωσης της ε, λειτουργίας του δικτύου με μια σειρά συστάσεων που προτίθεμαι να σας υποβάλω αγαπητοί συνάδελφοι. Το Solvit δημιουργήθηκε το 2002 από την Επιτροπή, ε, κατόπιν πρωτοβουλίας Επιτροπής ε, και θέλει να επιλύσει τα προβλήματα που ενδεχομένω αντιμετωπίζουν οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις λόγω ανεπαρκούς ε, αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εσωτερική αγορά. Το Solvit είναι σημαντικό γιατί παρέχει υποστήριξη για τους ε, πολίτες που καμιά φορά πρέπει να παλέψουν σκληρά για να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς. Πολλές φορές οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται ταχείες λύσεις και δεν ε, χρειάζεται να χάνουν το χρόνο τους ε, μέσω δικαστικών διαδικασιών. Γι' αυτό το Solvit συστάθηκε για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Ε, δεν παρέχει μόνο κάποιες λύσεις σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά είναι βασικός παράγοντας για την πρόληψη προβλημάτων που ενδεχομένως ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των κανόνων της ε, κοινή αγοράς εκ μέρους των χωρών μελών. Καμία φορά χρειάζεται αναθεώρηση του εθνικού, της εθνικής ή των μέτρων εφαρμογής. Ε, τώρα, υπάρχουν ε, κάποιες προσφυγές από τις διοικήσεις των χωρών μελών αλλά πολλές φορές προλαμβάνουν αυτές τις περιπτώσεις μέσω διορθωτικών μέτρων. Εάν δούμε τώρα τα στοιχεία, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι Solvit είναι πραγματική επιτυχία. Το 2008 υπήρχε αύξηση της τάξης του 22% των περιπτώσεων. Πάνω από χίλιες περιπτώσεις 83 ε, από αυτές ε, επιλήθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο, κάτι που είναι ιδιαίτερο συμφερεντικό. Αυτό μας δείχνει ότι το Solvit πραγματικά έχει την εμπιστοσύνη του πολίτη και των επιχειρήσεων. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο αξιοπιστίας για το δίκτυο αυτό. Παρ' όλα αυτά το Solvit έχει περιθώρια βελτίωσης. Υπάρχουν ορισμένε δυσκολίε που θα ήθελα να τις εξετάσουμε από κοινού και τις οποίες εγώ πρότεινα ορισμένες ε, βελτιώσεις στο σχέδιο έκθεσης και βεβαίως αναμένω πολλές άλλε προτάσεις προτάσεις υπό τη μορφή τροπολογιών. Καταρχήν θα ήθελα να πω κάτι το οποίο ήδη υπόθηκε. Υπάρχει έλλειψη επαγρύπνησης εκ μέρους των ε, ε συνειδητοποίηση εκ μέρου των πολιτών όσον αφορά την ύπαρξη του Solvit. Πολλέ φορέ οι πολίτε αγνοούν την ύπαρξη του Solvit και αγνοούν τι δυνατότητε που έχουν στη διάθεσή του για να επιλύσουν ε, τάχιστα τα προβλήματα που ανακύπτουν στην εσωτερική αγορά. 800.000 ευρώ, 1 εκατομμύριο ή ένα εκατομμύριο ευρώ, εάν τα πάρουμε τον επόμενο χρόνο, δεν είναι αρκετά. Παρ' όλα αυτά, είναι καλά για να οργανωθούν μεγάλες ενημερωτικές εκστρατείες. Ε, ε θα ήθελα να καλέσω τι χώρε μέλη να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι η εκστρατεία αυτή θα πρέπει να έχει πιο ποιοτικό χαρακτήρα, εξηγώντα επακριβώ τι μπορεί να κάνει το Solvit. Δεν περιμένουμε να δούμε σε αυτοκινητοδρόμους ε, ταμπέλες του τύπου εάν έχετε ένα πρόβλημα το Solvit θα σας το λύσει. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο σημαντικό πρόβλημα, το πρόβλημα ε, των ανθρώπων που απασχολούνται για να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό ε, χρειαζόμαστε περισσότερε πληροφορίε για τον πολίτη και τι επιχειρήσει, αλλά αυτέ οι, επιχει... πληροφορίες θα πρέπει να είναι εστιασμένε και θα πρέπει να εξηγούν ξεκάθαρα ε, ποιο είναι ο σκοπό του Solvit. Γιατί το Solvit έχει πέσει ήδη θύμα τη ίδια τη επιτυχία Σε ορισμένε ε, χώρε είναι υπερβολικά φορτωμένο Γι' αυτό θα πρέπει να αυξηθούν ε, τα κέντρα αυτά λαμβάνοντας ε, υπόψη τις περιπτώσεις που έχουν επιληθεί αναχώρα από το Solvit στο παρελθόν. Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη υπάρξει συγγνώμη, μεγαλύτερη σεβαστοποίηση για το Solvit μπορεί να αυξήσει αυτό το φόρτο. Ε, και αν αυξηθούν οι περιπτώσεις προσφυγής στο Solvit, πιθανόν να μειωθεί η αποτελεσματικότητά του. Προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να είναι το εργαλείο μέσω του οποίου να διανέμονται οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του Solvit, και με αυτό κλείνω την παρουσίασή μου, Χρειάζεται επίσης να οργανώσουμε επαρκές πρόγραμμα κατάρτισης των υπαλλήλων που εργάζονται στο πλαίσιο του Solvit, καθώς και εκείνων που απασχολούνται ε, στις διάφορες υπηρεσίες της ε, κυβέρνησης, ε, αλλά και να βελτιωθεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες ε, που ασχολούνται με νομικά θέματα. Γιατί πολλές φορές ε, τα ζητήματα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και πραγματικά χρειάζεται μια υποστήριξη όσον αφορά τα νομικά ζητήματα. Αυτή η βοήθεια μπορεί να έρθει από τις διάφορες ε, διοικητικές υπηρεσίες αλλά και από τις Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο της Επιτροπής για όλες τις ε, πληροφορίες ε, που μας παρήχε και την συνεργασία ε, σε σχέση με την έκθεση αυτή. Επίσης τον Τζόναθ Παπ από τη Γραμματεία της δικής μας Επιτροπής. Θα ήθελα η έκθεση αυτή πραγματικά να είναι θετική, γιατί το Solvit είναι ένα δίκτυο το οποίο νομίζω οφείλουμε να ολοκληρώσουμε να αξιοποιήσουμε την αποτελεσματικότητά του, η οποία μέχρι τώρα ήταν πραγματικά σημαντική, και να βρεθούν και δυνατότητες ε, αύξησης της αποτελεσματικότητας αυτής μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πουσόη. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια ιδιαίτερως περιεκτική παρουσίαση του θέματος αυτού. Και τώρα θα ακούσουμε τους εισηγητές, την κυρία Άνσλε, εκ μέρους της κυρίας Ρόιτεβα. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Ρόιτοβα δεν μπορεί να έρθει σε αυτή τη συνεδρία της Επιτροπής γιατί βρίσκεται σε μία ε, αντιπροσωπεία και στην Αφρική. Γι' αυτό εν ονόματι της θέλω να παρουσιάσω διάφορα από τα σχόλιά της. Ε, καταρχήν εν ονόματι της κυρίας Ρόιτοβα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που έχει καταρτήσει μία πολύ καλή έκθεση η οποία είναι ένα πολύ βασικό θέμα και συμφωνώ με όλα τα θέματα τα οποία έθεσε και ιδίως με αυτά τα οποία αναφέρονται στην ε, συνειδητο... καλύτερη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της ανάγκης προώθησης του θέματος αυτού, οργανώνοντας ε, την ε, επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων και των ε, συνδέσμων ε, σε εθνικό επίπεδο και στα Υπουργεία, την εμπλοκή του Κοινωνικού Ταμείου για να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα διαχειρήσεως του δικτύου εάν δεν υπάρχει επαλκές προσωπικό στα κέντρα Solvit. Και συμφωνώ επίσης ότι θα έπρεπε να τα στηρίξουμε τα θέματα αυτά. Το Solvit είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, οι οποίοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι έχουν ε, αντιληφθεί τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά, διότι πρόσφατες εκθέσεις αναφέρουν 83% των προβλημάτων που ελήφθησαν, δηλαδή ε, προβλήματα που έθεσαν οι πολίτες και συμβουλές που έλαβαν οι πολίτες. Σύμφωνα με την κυρία ε, Ρόιτοβα πρέπει να αυξήσουμε την προβολή του συστήματος αυτού για να αναγνωρίζεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η εκστρατείες που θα εστιάζονται σε ορισμένους αποδέκτες θα πρέπει να οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων. Επίσης, ε, η εσωτερική αγορά ε, πρέπει ε, να ολοκληρωθεί με συμμετοχή του Solvit και στις περισσότερες περιπτώσεις όταν χρησιμοποιούμε το Solvit αναφερόμαστε σε ε, πολίτες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τα κοινωνικά τους δικαιώματα ή την αναγνώριση των επαγγελματικών τους διπλωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα με, σε συνεργασία με τις ενώσεις των αποδήμων ε, και με τα προξενία τα, στα οποία απευθύνονται οι ε, ενδιαφερόμενοι για να ζητήσουν πληροφορίες. Να βελτιώσει κανείς και την πρόσβαση στο Solvit μέσω του διαδικτύου. Διότι αν ένα άτομο ή ε, μία εταιρεία ε, γράψει την ε, διεύθυνση της ιστοσελίδας www.solvit.eu ή άλλες παραλλαγές ε, δεν ε, πρόκειται να καταλήξει στη σελίδα του Solvit. Πρέπει να γνωρίζει όλη την σελίδα ε, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή να μπει στο Solvit μέσω του Google η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να λάβει περισσότερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ε, επόμενη ε, έκθεση διότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να κληθούν μεμονωμένα και δεν μπορούμε να προτείνουμε λύσεις για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά τους. Ο καθένας έχει σωστές ε, επαφές με τα κράτη-μέλη και ε, πρέπει να ε, μπορέσουμε να επηρεάσουμε καλύτερα το θέμα αυτό σε συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών που πρέπει να ενισχυθεί. Όσον αφορά τη συμμετοχή στο ΚΟΖΑΚ, που είναι ε, μια επιτροπή που ασχολείται με τις ε, ε, με τις διάφορες ενώσεις θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εν ονόματι της κυρίας Ρόιτοβα να συγχαρώ και πάλι τον εισηγητή και να το πω ότι συμφωνώ με τα σχόλιά του. Όντως είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, απλούστατα δεν μπορούμε να το αξιοποιήσουμε όσο χρειάζεται. Ευχαριστώ για τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά σχόλια τα οποία θα βοηθήσουν τον εισηγητή να ολοκληρώσει τον κατάλογό του η κυρία Στάιλερ. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή ε, και ε, την εκπρόσωπο της κυρίας Ρόιτοβα για τα σχόλιά της. Εάν όμως λάβετε υπόψη σας ότι Ε, υπάρχει κάποια ανταπόκριση, θεωρούμε ορισμένα πράγματα δεδομένα. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε εντός του Κοινοβουλίου να ε, αναλάβουμε δράση, να εξτάσουμε το τι γίνεται στα κράτη-μέλη, διότι έχετε πληροφόρηση, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο στην εσωτερική αγορά και πρέπει ε, να εξασφαλίσουμε ότι τα πράγματα πάνε καλά, διότι διαφορετικά ε, όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα βλέπουμε ότι η εσωτερική αγορά ε, πρέπει ε, να λειτουργεί χωρίς να καταφεύγουμε εις, ε, εις τα δικαστήρια ε, και συμφωνώ με την άποψή σας διότι ε, ε, όταν χρησιμοποιούμε στο Ηνωμένο Βασίλειο το Solvit και αυτό το είπαν και οι προλαλήσοντες διαπιστώνουμε ότι πρέπει να ενημερωθούν περισσότεροι ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκεί πρέπει να εστιαστείτε να προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε διότι δεν το γνωρίζουν όλοι και επανέρχομαι εδώ στην προηγούμενη συζήτηση την οποία έπρεπε να, εξε... να λάβουμε υπόψη. Όσον αφορά τα οριζόντια προβλήματα, συμφωνώ και εγώ και όσον αφορά τα μέτρα τα οποία προβλέπετε είναι ενδιαφέροντα. Θα πρέπει και αυτό ίσως να το εξετάσουμε, τις ανταλλαγές των βελτίστων πρακτικών, τι μπορεί να λειτουργήσει στα διάφορα κράτη, διότι πολλές φορές το θέμα του προϋπολογισμού είναι ενδιαφέρον, αλλά όπως έχουμε πει και στο παρελθόν θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα, να δούμε γιατί δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και από εκεί να ξεκινήσουμε να δούμε πώς πληρώνουν το προσωπικό τους και ε, επίσης το θέμα της δημοσίευσης, το θέμα της πληροφόρησης. Πρέπει να, όλα αυτά να τα κοιτάξουμε από δύο διαφορετικές σκοπιές, γιατί αναφερθήκατε εις ε, την ε, ηλεκτρονική πύλη, στο διαδίκτυο, Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα και δεν θέλουμε ε, να καταπολεμήσουμε την επάνδρωση με προσωπικό. Απλούστατα πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε όταν ζητάμε περισσότερους πόρους για ενημέρωση του κοινού και ε, για προσωπικό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται με την νομοθεσία η οποία έχει παρανοηθεί διαμέσου των ετών και στην ε, εξαρτή ενημέρωση όλοι είπαν ότι πρέπει να καταστούμε πιο αποτελεσματικοί. Οπότε ε, θα πρέπει ίσως να εστιαστούμε σε εκστρατείες που θα οργανώνονται επιτόπου τόπου ε, και να καθορίζουμε προθεσμίες. Έτσι, εάν κάποιος αναλάβει ε, ένα θέμα που είναι εκτός της εντολής του ε, για να ε, προωθήσει το Solvit θα πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται γιατί ίσως είναι δυνατόν να λειτουργήσουν διαδικασίες που δεν έχουν άμεση σχέση με το Solvit και εκτός του Solvit Είμαστε όμως 750 και ευρωβουλευτές και θέλουμε να προσπαθήσουμε ε, τους πολίτες και τους καταναλωτές σε κάθε χώρα. Ευχαριστώ την κυρία Στάιλερ, συμφωνώ ε, με το θέμα αυτό που πρέπει να συζητήσουμε ε, με ε, το, τους νέους επιτρόπους. Είχαμε υποβάλει το θέμα στον κύριο Μακρύβη πριν από κανένα εξάμηνο αλλά καλό θα ήταν οι νέοι επίτροποι να μπορέσουν εγκαίρως να επέμβουν και να χρησιμοποιήσουν τη δικιά τους μέθοδο. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να προτείνω πολλά γιατί υπήρξαν και τα σχόλια της κυρίας Χάσλικ αλλά αναφέρουμε εδώ στην ιστοσελίδα, στην προβολή συμφωνώ με τα σχόλια της κυρίας Στάιλερ και καλό θα ήταν να ενημερώσουμε τους νέους ευρωβουλευτές γιατί και εγώ όταν ε, έχω ερωτήματα από τους πολίτες και τους παραπέμπω στο Σόλβι, τους κάνει καλό το οποίο πρέπει να γίνει και με τους νέους ε, ευρωβουλευτές για να μπορούν να διοχετεύουν στη σωστή κατεύθυνση τα ερωτήματα ε, των ε, των ψηφοφόρων τους αν έχουμε χρησιμοποιήσει το σωστό τρόπο για τη χρηματοδότηση είναι κάτι που με προβληματίζει διότι έχω ορισμένε ερωτήσεις και πιστεύω ότι του θέματος αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μας λύσει το πρόβλημα. Ο κύριος Τερκούσκι. ήθελα να μιλήσω πολωνικά. Υποστηρίζω την έκθεση, η οποία πραγματικά είναι πολύ, έχει, πολύ καλογραμμένη. Νομίζουμε ότι μπορούμε να δούμε πόσο σημαντικό είναι το Solvit όταν μιλάμε για τον προπολογισμό και τις περισσότερες φορές συζητάμε κατ' ουσία για το Solvit. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μπουσόη που μας έφερε τα ευχάριστα νέα για την αύξηση του προϋπολογισμού από 800.000 σε 1 εκατομμύριο ευρώ. Ακούσαμε την άποψη εδώ, το Solvit έχει πέσει θύμα της ίδιας της επιτυχίας και όλο και... και ότι δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό Γι' αυτό υπήρξαν κάποια παράπονα το 2007 γιατί οι διαδικασίε ήταν τόσο ταχείε. Το 2007 ήταν 85 μέρες. Και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό που η έκθεση αναφέρει την διάθεση να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του Solvit ε, με, μέσω της ενίσχυσής του από, με περισσότερα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πραγματικά με θεώρησα την ενδιαφέρον ότι κάθε χρόνο υπάρχει μια αύξηση των παραπάνω εκ μέρους των πολιτών. Αλλά από την άλλη, ο ρυθμός των επιχειρήσεων που προσφεύγουν στο Solvit ε, παραμένει χαμηλός. Ε, και νομίζω ότι θα έπρεπε τα μέλη του Solvit να παράσχουν τη συνδρομή τους στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να εξετάσουμε το φαινόμενο αυτό, ούτως ώστε να θεσπίσουμε κάποιες ε, κατευθυντήριες γραμμές για να προαγάγουμε το Solvit περισσότερο μεταξύ των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που επεσήμανε η κυρία Κέπερτ. Εγώ άκουσα πρώτη φορά για το Solvit όταν έγινα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρόλο που ήμουν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Πολωνικού Κοινοβουλίου ε, και εγώ η ίδια υπήρξε επιχειρηματίας, αλλά ε, ποτέ δεν είχα ακούσει για το Solvit, μόνο όταν έλαβα το έργο αυτό η συγκίτρια Είναι παράδοξο λοιπόν το γεγονός ότι ενώ το ίντερνετ είναι το βασικό μέσο για την ύπαρξη του Solvit, το ίδιο το Solvit αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα με το ίντερνετ. Η κυρία Χέντρι το ανέφερε αυτό. Το Solvit δεν έχει ένα συντονισμένο σύστημα εθνικών ιστοσελίδων. Το έλεγξα σήμερα πριν από αυτή τη συνεδρίαση και διαπίστωσα ε, ότι οι, διευθύνσεις των, οι εθνικές διευθύνσεις του Solvit ε, έχουν εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους περιεχόμενα. Το Solvit ε, θεωρείται, η ύπαρξη Solvit θεωρείται αυτονόητη, ωστόσο δεν χρησιμοποιείται συχνά μέσω του ίντερνετ. Η C, Europa.solvit. Είναι η διεύθυνση Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή άμεσα, αν δεν έχουμε τη σωστή διεύθυνση. Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου θα κατευθούν οι τροπολογίες. Εγώ ίδια έχω υποβάλει μια σχετική τροπολογία. Δηλαδή το Solvit είναι πραγματικά πολύ θετικό εργαλείο, αλλά προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του χρειαζόμαστε ε, περισσότερα κονδύλια και ένα streamlining ε, ε, νομίζω ότι έχετε δίκιο όταν λέτε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την ε, ευαισθητοποίηση των συναδέλφων στο επίπεδο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ όλους τους και συγητές. και τώρα έχω δύο άλλους ομιλητές στον κατάλογό μου. Την κυρία Βανιού πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσό για την εξαιρετική του εργασία. Νομίζω ότι έχουμε εδώ ένα ιδιαίτερο χρήσιμο εργαλείο που όπως υπογραμμίσατε όλοι δεν είναι ιδιαίτερο αποτελεσματικό. Θα πρέπει λοιπόν αν αυξήσουμε τα μέσα όταν μιλάμε για αποτελεσματικότητα των καταναλωτών και των πολιτών της Ευρώπης, αυτό είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καθημερινά. Και εγώ η ίδια έκανα το σχετικό έλεγχο, γιατί είχα πολλά προβλήματα που με υποβλήθησαν από τις πολίτες πριν από τις εκλογές και όπως κανείς δεν είναι αρμόδιος για όλα, τους παρέπεψα στο Solvit και συνειδητοποίησα ότι οι απαντήσει ήταν ε, εξαιρετικά ακριβεί σε εύλογε προθεσμίε. Και νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να κυκλοφορήσουμε την πληροφορία ότι το Solvit υπάρχει. Εγώ πήρα κάποια φυλάδια ενημερωτικά, τα έβαλα στη μαρχία κλπ. Και συνειδητοποίησα ότι πράγματι υπήρχε ζήτηση αλλά και μια απόκριση εκ μέρους του Solvit. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει ένα προϋπολογισμό. Γιατί είναι δυνατόν να παράσχονται αυτές οι πληροφορίες, αλλά αυτό προϋποθέτει ένα επιπλέον προϋπολογισμό με κανόνα ικανούς ανθρώπινους πόρους. Και βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια δημόσια ενημέρωση σε όλους τους δημόσιους χώρους. Και έτσι οι πολίτες θα κατανοήσουν πόσο η Ευρώπη μπορεί να εισβάλλει στη βελτίωση της καθημερινής του ζωής. Είμαι σύμφωνη με την κυρία Ρούλ. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν είναι το ενδεδειγμένο όργανο χρηματοδότησης γιατί ε, δεν επαρκή. Ε, χρησιμοποιείται πάρα πολύ για θέματα εδαφικής συνοχής. Χρειάζεται ένας ειδικό προϋπολογισμός στο ύψος των δικών μας στόχων και φιλοδοξιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, σημείωσα τις παρατηρήσεις σας ιδιαίτερα για την διαστημότητα του Solvit στη Γαλλία. Ε, και πραγματικά θα ήθελα να αναγνωρίσω το γεγονός, να χαιρετήσω το γεγονός ότι ο μόνος αντιπρόσωπος εθνικής κυβέρνησης είναι από τη Γαλλία. Ε, και πραγματικά υπάρχει μεγάλο ζήλος για το Solvit στη Γαλλία θα, θα ακούσα τις παρατηρήσεις της κυρίας Βανιού για την ε, διαθεσιμότητα του Σόλβιτ στη Γαλλία. Κύριε Γκρέγκ, έχετε το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο γιατί τέθηκαν, ε, καλέθηκαν πάρα πολλά σημεία από του προηγούμενου ομιλητέ. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσό για την έκθεσή του. Παρ' όλα αυτά, έχω μια σύγχυση. Είπαμε ότι έχουμε στεσμένε πληροφορίε. Ε, ε, όταν, αλλά λέμε από την άλλη ότι δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες. Είπατε επίσης ότι το Solve ήταν πετυχημένο σε όλες τις χώρες μέλη. Θα ήθελα να έχω κάποιες πληροφορίες κατά πώς τα ποστά αυτά επιτυχίες κατανέμονται ισομερώς σε όλες τις χώρες και αν όχι γιατί. Τώρα, όσον αφορά την κατάρτιση, Προφανώς αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι όταν αναφέρουμε μια γραμμή του προπολογισμού, είπαμε ότι αρχικά ήταν 800.000, τώρα είναι εκατομμύριο ευρώ. Ε, ξέρουμε πως θα χρειαζόμαστε, γιατί το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δεν είναι πραγματικά μια εναλλακτική λύση. Θα πρέπει για το 2011, προκειμένου να υπάρξει επιτυχία, χρειαζόμαστε 1,2. Και αυτό είναι το ειδικό ποσό που χρειαζόμαστε προκειμένου το εργαλείο αυτό να, αποβεί, να στεφθεί με επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, θα συνεχίσω στα δανικά, δανέζικα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση του κυρίου Μπουσό είναι ιδιαίτερος πετυχημένη και όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ε, νομίζω ότι εδώ το θέμα δεν είναι τόσο τα χρήματα κονδύλια, αλλά οι εμπειρίες που υπάρχουν στα διάφορα κέντρα Solvit. Ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια, ένα είδος ακρόαση στις διάφορες χώρες μέλη, στα διάφορα κέντρα, για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες τους και τι επιδέχεται βελτιώσεων στη βάση της υπάρχουσας εμπειρίας. Και βεβαίως εδώ θα μπορούσε κανείς να εξετάσει το ενδεχόμενο να δοθούν, να υπάρξουν κάποια ερωτηματολόγια όσον αφορά την εμπειρία μέχρι τώρα. Γιατί οι εμπειρίε αυτές μπορεί να είναι διαφορετικέ από τη μία χώρα στην άλλη. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε αυτή τη μικρή έρευνα γιατί όπως είπαν και οι προηγούμενες ομιλητές, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το Solvit, το θέμα δεν είναι μόνο τα χρήματα, αλλά να αξιολογήσουμε την εμπειρία μας μέχρι τώρα. Αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο, πιστεύω. Να ευχαριστήσω όλους για την ε, αξιόλογη φορά τους Και τώρα θα ήθελα να καλέσω την κυρία Γκρούμπερ εκ μέρους της Επιτροπής να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξάρω το έργο αυτής της Επιτροπής γιατί πραγματικά διαπίστωσε τα ωφέλη του Solvit ε, πριν από όλους. Όταν ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια με το Solvit, πολλοί εντός των θεσμικών οργάνων θεώρησαν ότι ε, ε, ότι δεν ήταν δυνατόν να ε, επιλύονται ε, τα, προβλήματα αυτά μέσω του Solvit σε μερικές εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ποιότητα των υπηρεσιών του Solvit, αλλά επίση και στην υποστήριξη αυτή τη επιτροπή καθώ και στην προβολή του Solvit, ιδέω εκ μέρου του κυρίου Χάρμπουρ, ο οποίο συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία του Solvit και ο οποίο και, και, και, καταφέραμε το Solvit μετά από αυτά τα 7 χρόνια να ε, καταστεί ορατό σαν ένα σημαντικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τώρα ε, ήταν κατάλληλη ώρα να συναχθεί αυτή η έκθεση ε, πρωτοβουλία σε σχέση με πολλά θέματα τα οποία διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα, ορισμένε γενικέ παρατηρήσει όσον αφορά αυτό το σημείο. Όσον αφορά την ε, περαιτέρω προώθηση του Solvit, συμφωνούμε ότι χρειάζεται μια τέτοια προώθηση, ιδιαίτερα όσον αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, γιατί αν δούμε τα στατιστικά δεδομένα, βλέπουμε ότι στερούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει όσον αφορά την προσφυγή του στο Solvit. Ωστόσο, Έχουμε παλέψει με αυτά τα ζητήματα προώθηση του Solvit τα περασμένα χρόνια και προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη προσέγγιση εδώ. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ε, μια έστω σόφρον ενημερωτική εξατία δεν θα βοηθήσει. Το 2007 ξεκινήσαμε το σχέδιο δράσης ενιαίας αγοράς, το οποίο θα σας παρουσιαστεί πιο λεπτομεριακά τον Ιανουάριο, αν δεν απατώμε. Αλλά θα ήθελα να κάνω τώρα μερικέ παρατηρήσει όσον αφορά τη διασύνδεση μεταξύ Solvit και αυτού του προγράμματο δράση. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε στο πρόγραμμα δράση είναι να προαγάγουμε όχι μόνο το Solvit, αλλά όλο το πακέτο υπηρεσιών που έχουμε στη διάθεσή μα. Γιατί για να πάρουμε ένα παράδειγμα, θα έλεγα το εξή, το Solvit ε, έχει σαν σκοπό να ασχοληθεί με συγκεκριμένα προβλήματα. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν ε, αντιμετωπίζουν μεν συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά έχουν γενικά έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά τις, ε, την νομική τους υποστήριξη για τα δικαιώματά τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχουν κάποιοι πάλι που θα μπορούσαν βεβαίως να απαντήσουν αυτά τα ερωτήματα. Πολλοί από αυτού απευθύνονται στο Solvit, αλλά το Solvit δεν είναι δεδομένο όργανο για να απαντήσει αυτά τα θέματα. Και οδηγεί αυτό το φαινόμενο σε κατασπατάληση χρόνου. Και νομίζω ότι θα ήταν πιο χρήσιμο αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι που να απαντούν αυτά τα ερωτήματα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια συνδυασμένη προσπάθεια προώθησης ε, δηλαδή ε, τις υπηρεσίες ενημέρωσης των ε, πολιτών εν γέννη. Όχι όμως με διαφορετικές ταμπέλες, γιατί αυτό προκαλεί σύγχυση. Γιατί η πείρη μας είναι ότι οι άνθρωποι θα βρουν το δρόμο τους στο Σόλβιτ όταν το χρειαστούν ειδικά. Αυτό που χρειάζεται να μπορούν να κάνουν είναι να βρίσκουν το Solvit μέσω του Google, μέσω του Ιντερνετ. Γι' αυτό οι παρατηρήσει σα σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων και τη δυνατότητα να βρίσκεται το Solvit μέσω του Ιντερνετ είναι απολύτω ε, ουσιαστικέ. Και θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε την ιστοσελίδα του Solvit, ούτω ώστε αν κάποιο, για παράδειγμα, αναφέρει έχω πρόβλημα με, ε, με την άδεια οδήγηση, να μπορούν μέσω του Google να προσφύγουν στην περίπτωση αυτή στο Solvit. 70% των περιπτώσεων ε, που προσέφηκαν στο Solvit το 2009 δεν ε, απευθύνθηκαν στο κατάλληλο εργαλείο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών. Πέρσι εφαρμόσαμε ε, μια κοινή online υπηρεσία ε, συστήσαμε μια κοινή online υπηρεσία, ένα κοινό σημείο πρόσβασης ε, που τους κατευθύνει ανάλογα, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Και αυτό είναι ένα σύστημα που θέλουμε να επεκτείνουμε και σε άλλες υπηρεσίες. Γιατί ε, οι πολίτες, όπως είπατε, χρειάζεται να ξέρουν τα ονόματα όλων αυτών των επιμέρους υπηρεσιών. Τώρα, ένα άλλο θέμα. Στο σχέδιο έκθεσης ο εισηγητής αναφέρει τη χρησιμότητα συστημάτων όπως το Solvit ε, σε σχέση με προβλήματα στην εσωτερική αγορά. Αυτό το αναγνωρίζουμε στο πρόγραμμα δράση της εσωτερικής αγοράς για το Solvit και οι άλλες υπηρεσίες έχουν ε, ιδιαίτερα χρήσιμο feedback ε, για την Επιτροπή και το Συμβούλιο εν σχέση με το τι λειτουργεί στην ιστορική αγορά και τι δεν λειτουργεί. Και επίσης μπορούμε να μας πούν ε, σε ποιους ε, τομείς οι πολίτες χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά τους. Ένα πρόγραμμα λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε ε, να παράγουμε κάποιες εκθέσεις σε σχέση με την ενιαία αγορά σε τήσια βάζη. Και το 2011 θα βαστεί η έκθεση αυτή σε <coughs> περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του Solvit αλλά και των κέντρων Ευρωπαίων καταναλωτών. Αυτό είναι μεγάλο έργο για μας γιατί πρέπει να συνεργαστούμε με όλες τις ε, ενεχόμενες υπηρεσίες αλλά από την άλλη θα έχουμε μια ε, πλήρη εικόνα σχέση με τι συμβαίνει στην εσωτερική αγορά και με το πώς οι πολίτες προσλαμβάνουν την εσωτερική αγορά όσον αφορά τις ε, αγορές που κάνουν αλλά και τα προβλήματα που έχουν με τις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες. Αυτό είναι το πρόγραμμα λοιπόν για το 2011. Τώρα, ένα από τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα με το Solvit είναι το προσωπικό. Και πολύ αναφερθήκατε σε αυτό το θέμα. Η εικόνα είναι λίγο μεικτή εδώ, γιατί αν δούμε τα στοιχεία της έκθεσης του περασμένου χρόνου και του φετινού, που θα βγει σε λίγο, ε, θα δείτε ότι ε, οι χώρες μέλη έκαναν μέχρι στιγμής αρκετά πράγματα για να αυξήσουν το προσωπικό, αλλά υπάρχουν άλλες χώρες όπου το προσωπικό είναι ιδιαίτερως ισχνό και χαίρομαι πια από αυτές τις μεγάλες ε, χώρες που παρίσταται εδώ γιατί εκεί ε, το Solvit το προσωπικό αποτελείται από σταζιέρ ε, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι ε, πολύ καλό για την χώρα αυτή. Στο σχέδιο έκθεσης υποδεικνύεται το ενδεχόμενο να εισφέρει το κοινωνικό ταμείο στα ζητήματα προσωπικού. Αλλά όπως κυρία Ρούλη έχουμε φουλής κατά πόσο αυτό μπορεί να δουλέψει γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν έχει σαν σκοπό να προσλαμβάνει εθνικούς υπαλλήλους. Ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στις χώρες σύγκλησης, αλλά όχι στις μεγάλες χώρες και έχουμε σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Τώρα, μία άλλη πρόταση έγινε από την κυρία Χάμσλινγκ, αν δεν απατώμε, που είναι πιο ενδιαφέρουσα για εσά, του βουλευτέ, ω υπέρμαχα του Σόλβιτ να επικεντρώσετε στι χώρε εκείνε όπου υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Αυτό είναι ο τύπο πίεση που είδαμε ότι αποφέρει αποτέλεσμα στο παρελθόν. Εάν λοιπόν μπορέσετε να δείτε ποιες είναι οι χώρες όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με το προσωπικό και μπορέσετε να σχεδιάσετε τη δική σας εκστρατεία για να βοηθήσετε και να πιέσετε, αυτό ενδεχομένω θα βοηθήσει τη βελτίωση τη κατάσταση με το προσωπικό. Γιατί η εμπειρία μου είναι όσο. Ε, ε, αυτή κανεί την πίεση, τόσο περισσότερα αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει. Τέλος, έγινε μια παρατήρηση σε σχέση με την οργάνωση μιας εκδήλωσης για τους βουλευτές. Συμφωνώ με την παρατήρηση αυτή, γιατί τα μέλη του Κοινοβουλίου είναι η πιο σημαντική μας υπέρμαχη την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά το Solvit. Ε, είμαστε στη διάθεσή σας για μια τέτοια διοργάνωση παρόλο που η διαφήμιση θα πρέπει να γίνει όχι μόνο για το Solvit, αλλά για όλες τις άλλες χρήσιμες υπηρεσίες ενημέρωσης του πολίτη που έχουμε στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Γκρούμπε για αυτή την πολύ περιεκτική σας παρουσίαση. Σημειώνομαι την σχετική έλλειψη προσωπικού στα κράτη-μέλη. Ίσως αυτό να είναι κάτι στο οποίο να θέλει να δώσει πρωτοβουλία. Και ξέρω ότι ο κύριος Μπαρνιέ είναι φοβερός χρήστης του Σόλβιτ, οπότε σίγουρα ένα σταζιέρ θα τον ε, απασχολεί μόνο γι' αυτό. Κύριε Μπουζόη, θέλετε να συνοψίσετε. Εγώ έχω ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω πως το έχετε κι εσείς. Πολύ σύντομα να πω κάποια πράγματα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που παρενέβησαν και που υπέβαλαν προτάσεις. Συμφωνώ με τα πέντε σημεία που έφερε η κυρία Χένσλικ στο όνομα της κυρίας Ρόιτοβα, αλλά και στο δικό της όνομα επίσης. Πιστεύω πραγματικά ότι οι μικρομεσαίες θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένες και αυτό είναι κάτι που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί να επιστήσω την προσοχή για το θέμα το ίντερνετ και του σχετικού site, κάτι που είπε και ο κύριος Κούρσκι. Και νομίζω πως θα πρέπει να εσωματώσουμε εδώ, στην έκθεσή μας, στην τροπολογία αυτή, πιο ξεκάθαρα site το ίντερνετ για το Solvit. Περισσότερη ενημέρωση για τα κέντρα Solvit επίσης συμφωνώ. ίσως στις αρχές της επόμενης χρονιάς με τον νέο επίτροπο. Σκέφτηκα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να είναι για το τοπικό ε, προσωπικό και ε, να απαντήσω και στον κύριο Γκρέχ και στη στην, κυρία Ρούλερ που ρώτησαν για τον προπολογισμό. 800.000 ευρώ ήταν ο προπολογισμό για το 2009. Ένα δις ήταν η πρότασή μας που υιοθετήθηκε και με τη δεύτερη ανάγνωση για το 2010. Αλλά αυτός είναι ο προπολογισμό για την προώθηση του Solvit και για την υπηρεσία για την ενιαία αγορά. Τα χρήματα αυτά δεν αρκούν για μεγάλη εκστρατεία ενημέρωση στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και ζητάμε από τα κράτη-μέλη να κάνουν ε, πολλαπλασιαστικέ δράσει, να χρησιμοποιήσουν τα ΜΜΕ για να προωθήσουν το Solvit. Τώρα, το προσωπικό. Αυτό το πληρώνουν τα κράτη-μέλη. Τα διάφορα υπουργεία, πληρώνονται λοιπόν από τα κρατημέλη και δουλεύουν μόνο για το δίκτυο του Solvit. Σε κάποιες χώρες έχουμε μόνο έναν άνθρωπο, ενώ σε κάποιες όλες έχουμε ανθρώπους που δεν μιλάνε αγγλικά για παράδειγμα. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο αριθμός των ανθρώπων που δουλεύουν για το Solvit, αλλά και η εκπαίδευση τους. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να ε, λύση. Είναι θέμα των κρατών μελών. Επίσης πιστεύω, και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση, ότι πέρα από το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μπορούμε να ακολουθήσουμε και την κυρία Βερνιό. Ο, κανένας μας, ο καθένας μας να οργανώσει στην περιοχή μας μια εκστρατεία ενημέρωσης για το τάδε δίνα μέσο και αυτό φυσικά θα βοηθήσει ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση για το Solvit. Το προχρονοδιάγραμμα το είχα ήδη προτείνει, παρουσιάσει μάλλον. Είμαστε τώρα στη 2 Δεκεμβρίου για την εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Είναι η πρώτη μου έκθεση, αλλά είναι και το, το γενέθλιο της συζύγου μου, οπότε η Δευτέρα Δεκεμβρίου είναι μια ιστορική ημερομηνία στο σταδιοδρομία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε 11 τη Δεκεμβρίου ως προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Παρακαλώ στείλτε λοιπόν τροπολογίες πριν την 11 Δεκεμβρίου. Η Επιτροπή ε, ε, Αναφορών θα υιοθετήσει την νομοδότησή της στις 23 Ιανουαρίου ε, και την έκθεση στις 8 Φεβρουαρίου ώστε να έχουμε πιθανότητες τον Μάρτιο στην πρώτη σύνοδο της Ολομέλειας να υιοθετηθεί η έκθεση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Δεν παρατήρησα ότι ήταν η πρώτη σας συνεδρίαση, η πρώτη σας μάλλον έκθεση. Συγχαρητήρια, όντως ιστορική ημερομηνία. Τελικό θέμα, για το οποίο έχουμε μισή ώρα, που ελπίζω θα είναι αρκετό για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Να καλωσορίσω τον Κλόντο Τούρμες εδώ, γιατί είναι μέλος της Επιτροπής μας και της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πασίγνωστος. Αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά που κάνουν έκθεση στην δική μας Επιτροπή. Η φήμη σου έχει ξεπεράσει και αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε μαζί μας εδώ. Και έχουμε επίσης και τον Φιλίπ Ζουβά. Εδώ. Η κύρια Παπανόβα δεν τη βλέπω εδώ. Έχετε μόνο δύο σκιώδεις εδώ σήμερα. Και νομίζω πως και ο υπεύθυνο τη είναι εδώ. Θα πάρει το λόγο αργότερα. Κλώτη Τούρμες, έχεις το λόγο για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και νομίζω πως θα μιλήσεις και για τις δύο προτάσεις από κοινού. Έτσι δεν είναι. Έχουμε την φαρμακοεπαγρύπνηση και την οδηγία και τον κανονισμό μαζί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ωραία να σου ρίχνω λουλούδια ακόμα για πριν να κάνεις οτιδήποτε. Ελπίζω να μην σας απογοητεύσω. Πρώτη μου εμφάνιση λοιπόν εδώ. Είναι τιμή μου να παρουσιάζω τις απόψεις μου για μια γνωμοδότηση. Καλημέρα στους και οδησηγητές. Νομίζω πως εμείς οι τρεις έχουμε ήδη πλειοψηφία. Οπότε αν συμφωνήσουμε ήδη από σήμερα, ήδη έχουμε προχωρήσει πολύ. Να παρουσιάσω τις ιδέες μου στα αγγλικά γιατί έπρεπε να ή να μπω στην ουσία του θέματος. Ο εμβολιασμός για την ε, για την κρύπη, το χειρό έδειξε ότι το κοινό δεν είχε μεγάλη ιδέα ότι βασικά όλες οι προσπάθειες να τους τραβήξουμε προς εμβολιασμό δεν λειτουργήσαν. Άρα λοιπόν πιστεύω πως αυτό το παράδειγμα δείχνει άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η οικοδόμηση εμπιστοσύνη. και βέβαια από πού πηγάζει η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη πηγάζει από την εμπιστοσύνη και τη γνώση της τεχνολογίας, από την διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών και ορισμένες φορές θα μπορούσε να αποτελεί και μια αντιφατική ανταλλαγή πληροφοριών, γιατί πολύ συχνά αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να πάρει κανείς, να έχει κανείς γρήγορα αποτελέσματα. Γνωρίζοντας ότι είμαστε μόνο μία από τις πολυάριθμες επιτροπές που εργάζονται με αυτό το ε, οδηγίες και τον κανονισμό, αυτό που έχω να προτείνω είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας να ε, επικεντρώσουμε την προσοχή σε θέματα που αφορούν τη δική μας Επιτροπή, δηλαδή τους πολίτες και την ενημέρωση των πληροφοριών και ε, να έχουμε όσο γίνεται πιο εναρμονισμένη προσέγγιση, ώστε να μην καταλήξουμε σε περιτούς φραγμούς στην εσωτερική αγορά. Εγώ θα εστιάσω σε δύο θέματα. Σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης που πρέπει να βελτιωθεί. Ενημέρωση για τα φάρμακα και τις φαρμακευτικές αγωγές και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε. Να σας πω ότι το γραφείο μου έχει κάνει κάποια έρευνα και υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ακόμα και για μένα ήταν εντυπωσιακά. Καταρχήν, η οι ε, νοσοκομιακέ νόσοι είναι η πέμπτη αιτία θανάτου αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν είναι καθόλου λίγο. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις Όπω α πούμε το Βάιοξ που μπήκε στην αγορά το 1996 για τη θεραπεία της γαστρίτιδας, ε, αποσύρθηκε το 2008 και τουλάχιστον σήμερα οι υπερογνώμονες λένε ότι αν είχαμε περισσότερη διαφάνεια για τις ε, παρενέργειες αυτού του φάρμακου, ορισμένοι άνθρωποι θα είχαν σωθεί. Και να μην πω και σε άλλα παραδείγματα. Η επαγρύπνηση λοιπόν θα πρέπει να αυξηθεί. Έχουμε θετικά παραδείγματα από την Δανία, τη Γαλλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, ε, την Ολλανδία, όπου υπάρχει περισσότερο ανοιχτό σύστημα και θα πρέπει να παρακινήσουμε όλους τους φορείς, τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς, τις φαρμακοβιομηχανίες, αλλά και τους πολίτες να έχουν μια πιο δραστήρια θέση, πιο δραστήριο ρόλο, ώστε να δίνουν πληροφορίες για αυτή, σε αυτήν την πλατφόρμα του ίντερνετ για τα επαγρύπνηση. Ορισμένοι λένε ότι πλημμυρίζουμε με πληροφορίες και έτσι τελικά δεν λειτουργεί το σύστημα, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που μπορούμε να λύσουμε να έχουμε αρκετούς πόρους ώστε να ταξινομήσουμε κάπως τις πληροφορίες. Αυτό που φαίνεται να είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι πως αυτό το σύστημα θα πρέπει να χρηματοδοτείται 100% από το κοινό, γιατί διαφορετικά θα έχουμε σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στους ε, προμηθευτές των φαρμάκων. Και δεν είναι ευχάριστο να βλέπουμε κάτι τέτοιο, να βλέπουμε παρατηρήσεις ή αμφισβητήσεις για τα ωφέλη. Όταν απειλείται η ζωή, νομίζω πως δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα για την εμπορική μυστικότητα. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως διαφανείς. Τώρα, ενημέρωση για τις ε, φαρμακευτικές αγωγές. Διάβασα κάποιο λόμπι που λέει ότι γιατί να μην πηγαίνει κανείς στο ίντερνετ, να, να, να ε, σώσουμε έτσι κάποια δέντρα και λίγο κόστος, γιατί ναι, είναι πολύ το χαρτί για τα φάρμακα και θα μπορούσε να μειωθεί. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουμε καταρχήν ότι αυτά οι πληροφορίες, τα PIL, δηλαδή οι πληροφορίες για τα φάρμακα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, είναι ήδη περιλήψεις. Τουλάχιστον το αν, ε, μου είπαν ότι αν αυτό περιοριστεί ακόμη περισσότερο δεν θα ήταν καλό γιατί κάθε σώμα είναι, είναι ξεχωριστό και δεν μπορούμε να περιορίζουμε υπερβολικά αυτές τις ε, πληροφορίες. Έπειτα το ίντερνετ καλό είναι, αλλά αν πάμε στις στατιστικές που ρωτάνε ποιο κομμάτι του πληθυσμού μας είναι ο μεγαλύτερος χρήστης ε, των ε, φαρμάκων, ακριβώς εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού που δεν ε, ασχολείται με το ίντερνετ. Πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Ορισμένοι από εμά είμαστε ενδιάμεσα σε κάποια κατηγορία ενδιάμεσα, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν και γραπτέ οι πληροφορίε. Τώρα για το θέμα του εμβολιασμού. Ε, πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί, ενώ υπάρχουν για τα 3, 4, 5 πρώτα χρόνια οι θετικές πληροφορίες, οι επιπλέον πληροφορίες για κάποιο φάρμακο, διαφορετικά όχι. Ε, γι' αυτό ίσως θα ήταν πολύ σημαντικό τα πρώτα χρόνια ο κόσμος να γνωρίζει πως πρόκειται για κάτι καινούριο, ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επιπλέον πληροφορίες γι' αυτό, εφόσον είναι νέο το φάρμακο ή το εμβόλιο. Αυτά Νομίζω πως αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας ως ΣΥΝΚΟ, γιατί έτσι θα έχουμε και μεγαλύτερη αξιοπιστία με τους υπολείπους. Uh, uh, Ευχαριστώ για τις πολύ σαφείς ε, εξηγήσεις σου και συμφωνώ ότι θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί ε, όταν θα έχουμε ένα σαφέστερο πλαίσιο. Και οι σκιώδεις φαντάζομαι θα συμφωνήσουν και δίνει το λόγο τώρα στον κύριο Ζουβά που είναι σκιώδης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο σε αυτή την ιστορική ημέρα, διότι όπως ξέρετε η 2 Δεκεμβρίου είναι για τη Γαλλία, για τη γαλλική ιστορία μια σημαντική ημερομηνία, διότι ε, σαν Βρετανός ίσως θα το εκτιμήσετε είναι η ημερομηνία της τέψεως του Ναπολέοντα του πρώτου. Στο θέμα της φαρμακοεπαγρύπνησης θέλω να κάνω μια γενική παρατήρηση και μετά δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Καταρχήν είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα τα φάρμακα είναι όλο και πιο αποτελεσματικά. Άρα δημιουργούν όλο και περισσότερες παρενέργειες. Τα φάρμακα που δεν έχουν παρενέργειες συνήθως δεν είναι πολύ χρήσιμα και είναι ίδιον ε, της ε, όλο και ε, πιο αποτελεσματικής αλλά και προϊούσης ιατρικής να δημιουργεί προβλήματα. Είναι άλλωστε αληθές ότι δεν έχουμε πολλούς ικανοποιητικούς αριθμούς και γιατί και επανέρχομαι γιατί ένα από τα χαρακτηριστικά της ε, παθολογίας η οποία οφείλεται εις ε, την ε, ιατρική αγωγή και αυτό είναι και το, το θέμα με τα φάρμακα οφείλεται σε μία έλλειψη δηλώσεως των ατυχημάτων. Επίσης ε, ε, τα φάρμακα επηρεάζουν και την νοσοκομιακή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Βέβαια μπορεί να πεθάνει κανείς ε, στο νοσοκομείο από πολλά πράγματα και συνήθως οι άνθρωποι πλέον δεν πεθαίνουν σπίτια τους αλλά στο νοσοκομείο ατυχώς και πολλές φορές από παρενέργειες φαρμάκων, παθολογικές παρενέργειες και από επιπτώσεις των ε, χειρουργικών επεμβάσεων και ούτω καθεξής. Άρα ε, το ουσιαστικό θέμα είναι το θέμα του γιατί σήμερα η φαρμακοεποπτεία δεν λειτουργεί σωστά. Θα είχαμε άδειο λοιπόν στην Επιτροπή αυτή να μην εξετάσουμε αυτό το ουσιαστικό θέμα το οποίο σημαίνει ότι η φαρμακοεπιπτία δεν είναι αρκετά αποτελεσματική και υπάρχει μία ε, ε, ε, ανεπαρκής δήλωση. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε. Δεν θα έπρεπε για, κατά τη συζήτηση αυτή να θέσουμε το σωστό ερώτημα γιατί δεν δηλώνονται όλα τα περιστατικά. Εάν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε αυτή την έλλειψη επαρκών δηλώσεων, διότι διαφορετικά πιστεύω ότι δεν θα ανταποκριθούμε, θα προχωρήσουμε λιγάκι, αλλά αυτά που θα επιτύχουμε δεν θα επαρκούν. Ε, χρειάζονται δηλαδή νέα στοιχεία και από το νέο στοιχείο πρέπει να κάνουμε προτάσεις. Άλλοτε, προτάσεις. Άλλωστε η Επιτροπή μας ε, προσπαθεί να αυξήσει τις δηλώσεις των παρενεργειών και προτείνει στους ε, ε, ασθενείς να δηλώνουν μόνοι τους τις παρενέργειες. Βέβαια μπορεί να κατακλειστούμε από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα, θα διηγούνται ιστοριούλες που δεν έχουν καμία σχέση με τα φάρμακα και αυτό είναι προφανές. Διότι εγώ είμαι υπεύθυνο ε, για ένα, μια υπηρεσία πρώτων βοηθειών στο Παρίσι και ε, στην αλληλογραφία μου έχω, κατακλείζομαι από γράμματα για ανεπάρκεια Καλή καλών, ε, ε, ε, καλής νοσηλείας και δεν έχει καμία σχέση το αποτέλεσμα με αυτό που επικαλούνται. Πρέπει λοιπόν να μην δημιουργήσουμε διαδικαστικά κάποια αναταραχή. Ο εισηγητής είπε ότι θα επιθυμούσε η χρηματοδότηση να γίνει από τους δημόσιους πόρους. Συμφωνώ για ηθικούς λόγους. Αλλά συγχρόνως αναρωτιέμαι Στη Γαλλία εφέτος το έλλειμμα, το τρέχον έλλειμμα της ε, κοινωνικής ασφάλισης θα είναι γύρω στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν βλέπω λοιπόν τις δημόσιες υπηρεσίες να αποδεσμεύσουν επιπλέον πιστώσεις για την φαρμακοεποπτεία. Βέβαια είναι επιλογές, αλλά για την υγεία του κανείς κάνει πολλές επιλογές και όλοι οι ιατροί, όλοι οι ομάδες ασθενών θα εκφράσουν τις κατά προτεραιότητα επιλογές τους. Γι' αυτό να μην νομίζουμε ότι θα έρθει ο Άγιος Βασίλης και θα μας δώσει ε, ε, δημόσιους πόρους. Ε, εκεί υπάρχει μία μεγάλη ανησυχία. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή ε, υποέλεγχος να ενταχθούν και οι φαρμακοβιομήχανοι σε αυτή τη διαδικασία. Και τέλος, γενικά, οι προτάσεις σας είναι ενδιαφέρουσες γιατί εντάσσονται μέσα στην ιστορία, δηλαδή δίνουν περισσότερες ε, εξουσίες στους ασθενείς που ενδιαφέρονται για την υγεία τους και υπάρχει ένα σημείο τομή στην Ευρώπη μεταξύ των αγγλοσαξονικών χωρών όπου ο ασθενής έχει σημαντικό ρόλο στη λήψη της απόφασης και στις, λατινικές χώρες ε, όπως η Γαλλία όπου υπάρχει μία ητοπάθεια και δεν συμμετέχει ο ασθενής. Αλλά όλες αυτές οι κινήσεις συντονίζονται και όλο και περισσότερο ο ασθενής συμμετέχει στην απόφαση που τον αφορά. Και έχω πέντε συγκεκριμένα θέματα τώρα, τα οποία θα ήθελα να αναφέρω και τα οποία ίσως θα συζητήσουμε μεταξύ μας. Καταρχήν, την δημιουργία ενός θέματος επί των πληροφοριών του φαρμάκου που δεν είναι καλή ιδέα γιατί δεν μπορούμε να συνοψίσουμε ουσιώδη πράγματα ε, να υπάρχει δημοκρατία βεβαίως είναι ουσιαστικό αλλά πρέπει μια πρώτη γνωμοδότηση να υπάρχει διότι επί 60 ημέρες οι άνθρωποι θα λένε ότι τους κατέβει και ε, πρέπει να μην δούμε μόνο τον κίνδυνο αλλά να αξιολογήσουμε τα υπέρ και τα κατά. Μετά, όσον αφορά τις ε, σοβαρές παρενέργειες θα πρέπει να αξιολογηθούν βάσει διεθνών προτύπων ε, στο τέταρτο σημείο συμφωνώ ότι πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε την περίληψη της περίληψης, όλα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και πέμπτον, θα ήθελα να υποφεληθώ από τις ερωτήσεις που δίθονται στην Επιτροπή για να ρωτήσω γιατί ε, δεν σταματάμε αυτή την τεχνική συνύπαρξη στον οργανισμό φαρμάκων μεταξύ της SHLP και ε, των άλλων οργανισμών διότι χρειάζεται αυτή η διητή ε, διάρθρωση και ίσως η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να σε εξηγήσει το ρόλο της Επιτροπής Συντονισμού και της SASP. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε με τις απόψεις σας. Και τώρα έχουμε 10 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Παβανόβα και μετά την κυρία Βάνιου θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ίσως θα ολοκληρώσει και το απόγευμα, αλλά εν πάση περιπτώσει η κυρία Παβανόβα έχει πρώτο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακόμη και αν δεν έχουμε συνεργαστεί ακόμη μαζί, ε, χαιρετίζω αυτή την ανταλλαγή απόφασης και πιστεύω θα συμφωνήσουμε σε πολλά θέματα, διότι εδώ το θέμα είναι πολύ βασικό για τους Ευρωπαίους ασθενείς και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και ανησυχίες. Αναγνωρίζω μεν και χαιρετίζω τον στόχο της ανασκευής των ήδη ενισχύ οδηγιών για να καταστούν πιο ορθολογιστικές. Αλλά όσον αφορά τα μέσα έχω αμφιβολίες ιδίως όσον αφορά την νομοτέλεια της ε, ε, χρηματοδοτήσεως από το δημόσιο των ε, κέντρων φαρμακο διότι νομίζω ότι αυτό δεν βοηθά να απεξαρτηθούν αυτά τα κέντρα από τις φαρμακευτικές εταιρείες και ίσως θα πρέπει να γίνουν επιλογές φορολογικές και δημοσιονομικές, ένα θέμα που θα συζητήσουμε μεταξύ μας και ε, αν ε, οι, οι φαρμακευτικές εταιρείες ελέγχουν την ερμηνεία των δεδομένων θα είναι εις βάρος των καταναλωτών. Δεν θα είναι ποτέ ανώδυνο και η άδεια της κυκλοφορίας πρέπει να γίνεται μετά από όλες τις αναγκαίες δοκιμασίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να γενικεύσει τα σχέδια διαχειρίσεως του κινδύνου που τώρα αναφέρονται μόνο στα πρωτότυπα φάρμακα ή στις εξαιρετικές διαδικασίες και όχι στα φάρμακα τα οποία θεωρούνται ότι είναι ισότιμα με ισχύοντα προϊόντα. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκε παραδείγματο χάρη για τα εμβόλια για την γρήπη Α χωρίς ε, να εμβαθύνουμε ε, και να εξετάσουμε τους ε, τρόπους παρασκευής και την δράση των προσθετικών στοιχείων. Αυτό βοήθησε τις φαρμακοβιομηχανίες, αλλά τώρα οι ασθενείς δεν είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα αυτά είναι ανώδυνα. Τι θα γίνει λοιπόν αν αυτή η μέθοδος γενικευθεί και οι ασθενείς, ε, βέβαια ε, το λέω πολύ σχηματικά, καθιστούν πειραματόζωα ε, μεγάλης κλίμακας και εκ των υστέρων μπορούν οι φαρμακοβιομηχανίες να διδαχτούν από τα λάθη τους. Πιστεύω λοιπόν ότι η ευρωπαϊκή βάση ε, είναι κάτι που μπορεί να μας ενδιαφέρει αλλά μας αφαιρεί όλη την ε, ειδική, όλο τον ειδικό χαρακτήρα των ε, φαρμακευτικών γνώσεων και πιστεύω ότι έτσι όπως προχωράμε θα αντιμετωπίσουμε πολλά, πολλές δυσκολίες διότι βάση δεδομένων δεν θα έπρεπε ε, να ε, ε, τροφοδοτείται παρά μόνο από τα εθνικά τις εθνικές βάσεις δεδομένων και μετά να δημοσιοποιείται. Θα πρέπει δηλαδή να εντείνουμε την ασφάλεια και την ε, εμπιστοσύνη όχι μόνο των ασθενών και των <clears throat> πολιτών αλλά και προς όφελος των φαρμακευτικών εταιριών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για αυτή την ε, πρόταση γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να μπορούμε να εμπιστευόμαστε τον, ένα τόσο σημαντικό τομέα της αγοράς όπως είναι ο τομέας των φαρμάκων. Θα ανατρέξω τα θέματα που ανέφεραν και οι συνάδελφοι όσον αφορά το σύστημα αναφοράς. Ε, ε, ε θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη, πιο αποτελεσματική φαρμακοβιομηχανία. Οι συζητήσει στο Συμβούλιο έδειξαν ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για το κατά πόσο η φαρμακοπαγρύπνηση είναι απολύτως αποτελεσματική στο πλαίσιο της οδηγίες. οδηγίας. Επιπρόσθετες απαιτήσει αναφέρονται στην έκθεση της Επιτροπής. Επιπλέον αναφορά ίσως θα πρέπει να αποφευθεί γιατί θα αυξήσει το φορτίο της ε, ε, των διοικητικών υπηρεσιών. Ε, όσον αφορά την αναφορά των ε, παρενεργειών, ε, εναπόκειται στους ασθενείς και έχει γίνει πολλές φορές, έχει υπάρξει άσκηση πίεσης εκ μέρους των ομάδων λόμπι των ασθενών. Ωστόσο, οι καταγραφή πληροφορίες πρέπει να είναι ευανάγνωστες για να εξυπηρεθούν οι στόχοι της φαρμακοπαγρύπνησης. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια όσον αφορά τις αναφορές εκ μέρους των ασθενών για τις παρενέργειες. Επίσης, όσον αφορά την επαρκή ενημέρωση όλων των είναι σημαντικό να ενημερώνονται έγκαιρα για τις ε, παρενέργειες, να τα αποτελέσματα ε, στη βάση μιας βάσης δεδομένων τους, ώστε να είναι άμεσα προσθέσει πληροφορίες. Γιατί πολλές φορές η φαρμακοβιομηχανία ε, είναι διατεθειμένη να αντιδράσει εφόσον ε, οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τις ε, εθνικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τα μέτρα σε σχέση με τις πληροφορίες που ε, δίδονται στους ασθενείς, νομίζω ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όταν μιλάμε για φάρμακα είναι ζωτική σημασία να έχουμε μια ισορροπία μεταξύ του κινδύνου και των, του φέλους του όφελου συγγνώμη, ενός φαρμάκου. Ε, γιατί οι ασθενείς θα πρέπει να αποτρέπονται χωρίς λόγο να, από τη χρήση του φαρμάκου και να διακόπτουν τη θεραπεία τους χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Ε, θα πρέπει, δεν θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο τις αποφάσεις χωρίς να συμβουλευθούν τον γιατρό τους. Όσον αφορά τώρα το ουσιώδες ε, με ιατρικούς όρους, σημαίνει δεν γνωρίζουμε, αλλιώς ουσιαστικό σημαίνει βασικό στην ε, κοινή γλώσσα. Δίνει λοιπόν ε, η διατύπωση αυτή λαβή σε παρανοήσεις και προτείνω να διαγραφεί αυτή η διατύπωση essential. Τώρα όσον αφορά ε, ειδική προειδοποίηση για ορισμένα προϊόντα ε, για προϊόντα τα οποία δεν παρακολουθούνται. Νομίζω ότι αυτό επίση δίνει λαβή σε αδικαιολόγητε ανησυχίε και κάνει του ασθενεί να σκέφτονται ότι υπάρχουν άλλα προϊόντα τα οποία παρακολουθούνται πιο αυστηρά. Τώρα, εάν αφορά τις, ε, όσον αφορά τις νέες πληροφορίες, να μπει αυτό σε εισαγωγικά, ε, να, μπει να γραφτεί με χαρακτήρες. Νομίζω ότι και αυτό δίνει λαβή σε παρανοήσεις. Τώρα, όσον... Ε, αφορά την οργάνωση της ε, διαβούλευσης με όλους τους ενεχόμενους. Ε, νομίζω ότι η έκθεση χαιρετίζει αυτή την ιδέα και καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για να υποστηρίξει αυτό το φυλάδιο της Επιτροπής που θα παράσχει εύληπτες και περιεκτικές πληροφορίες. Η εκθέση για την ασφάλεια του κοινού νομίζω θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ε, πανεπιστημιακών και ορισμένες από αυτές θα πρέπει επίσης να βρίσκονται στη διάθεση των ασθενών αντί να τους ε, παρέχονται πληροφορίες περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα που τελικά αυξάνουν την σύγχυση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τέρμες νομίζω ότι έχει ε, μια πολύ καλή ομάδα εμπειρογνωμόνων και είναι πολύ χρήσιμο που γίνεται η συζήτηση αυτή τη στιγμή γιατί όλα αυτά μπορούν να συμπεριληφθούν στο σχέδιο έκθεσής του. Ε, θέλετε να κάνετε κάποια εισαγωγικά σχόλια τώρα, θα έχετε την ευκαιρία να το κάνετε στο τέλος. Ε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσοι εξέφρασαν την ε, υποστήριξή τους. Θα ήθελα να περιστώ στο βασικό επιχείρημα της φαρμακοεπαγρύπνησης, δηλαδή την αύξηση της ε, διαφάνειας περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Θα πρέπει να σκεφτούμε, όπως υπόθηκε, ότι δεν περιλαμβάνει μόνο αναφορές στις περιπτώσεις ε, παρανέργειας των φαρμάκων. Ε, ο στόχος είναι μεν να υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά μπορεί να υπάρξει το αντίθετο αποτέλεσμα αν τα δεδομένα αυτά δεν είναι ανοιχτά στο κοινό. Τώρα, όσον αφορά την ε, ε, χρηματοδότηση ε, μπορεί να είναι εις βάρος του συστήματος μέσω επιβολής κάποιων τελών. Το σύστημα αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο, γιατί αυτή τη στιγμή το 75-80% ε, προέρχονται από αυτή την, των εισόδων προέρχονται από αυτή την πηγή και λιγότερο από 15% προέρχονται από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν πούμε λοιπόν τα χρήματα αυτά υπονομεύουν την αυτοτέλεια, ε, νομίζω ότι αυτή είναι μια δήλωση που σημαίνει ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο σύστημα συνολικά ως έχει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε την ε, εντύπωση ότι η βιομηχανία θα πρέπει επίσης να πληρώνει για την χορήγηση αδειών για τα φάρμακα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που διευκρινίζετε αυτά τα, θέματα. Ε, θέλετε να πείτε κάποια καταληκτικά λόγια. Εγώ πεινάω, το ίδιο και οι διερμηνείς. Έλαβα γνώση των προτάσεων, θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω όλα αυτά στην γνωμοδότησή μου. Νομίζω ότι χρειάζεται, ε, θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση των σκιωδών ε, αρχές Ιανουαρίου και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Ε, ίσως θα πρέπει να μοιραστούμε αυτό το φορτίο, το έργο. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, προτείνω να αποσταλεί το κείμενο